Chers collègues, je vais peut-être vous demander de bien vouloir prendre vos places. C'est le printemps. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έφτασε η άνοιξη, θέλουμε όλοι λίγο να ξεκουραστούμε και να δεν πελιάσουμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε, διότι είναι ιδιαίτερα φορτωμένη η σημερινή μας συνεδρίαση. Περιμένω να καθίσετε. Bien. Alors, tout d'abord, Προτείνω να περάσουμε στην έγκριση της μεσαίας διατάξεως. Η συνεδρίασή μου θα διαρκέσει σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Υπάρχουν διαφωνίες, ενστάσεις σχετικά με τη διάταξη. Όχι. Δεν έχω καμία ανακοίνωση να σας κάνω. Μόνο να σας πω ότι έχουν, διαθέτουμε όλες τις γλώσσες πλην ε, λετωνικών και εστονικών σήμερα στην συνεδρίαση. Δεν μπορώ να σας ζητήσω να εγκρίνετε τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 23 Φεβρουαρίου διότι δεν έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες ε, και έτσι αναβάλουμε την έγκριση των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης και φτάνουμε στο σημείο υποχρεώσει των φορέων εκμετάλλευση που διαθέτουν ξυλία και προϊόντα ξυλίας στην αγορά. Να σα υπενθυμίσω πω το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση ενέκρινε πρόταση κανονισμού στις 22 Απριλίου 2009. Το Συμβούλιο έχει μια θέση που είναι διαφορετική, είναι πιο εύκαμπτη, πιο χαλαρή θα λέγαμε από τη δική μας. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό και θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Καρολίν Λούκας. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κυρία Σέν, θέλει λάβει το λόγο. Α, συγγνώμη. Κυρία Λούκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχω σήμερα την ευκαιρία να τονίσω κάποια ζητήματα που με ενδιαφέρει να συμπεριφορική στη ανάγνωση. μερικά σχετικά με το ιστορικό. Όλοι γνωρίζετε ότι η παράνομη υλοτομία συνδέεται με μια σειρά προβλημάτων τόσο κοινωνικών όσο και περιβαλλοντικών. Οδηγεί στην αποδάσωση και συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της βιοποικιλότητας μειώνει τα έσοδα από την ε, φορολογία και αυξάνει την ε, φτώχεια των εξαρτωμένων από την υλοτομία. Νομίζω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να αναλάβει δράση κατά της ε, αποδάσωσης και της παράνομης ξύλευσης. Χρειάζεται λοιπόν να προστατεύσουμε την αγορά από την παράνομη ξυλία. Τώρα εμεί στην πρώτη ανάγνωσή μας ε, ενισχύσαμε ε, την πρόταση της Κομισιόν και συμπεριλάβαμε τις απαγορεύσεις στην ε, <coughs> εμπορία παράνομη ηλιοτομημένη ξυλίας και προϊόντος ξυλίας. Και θέλουμε να καλύψει αυτό όλους τους φορείς. Τώρα, το, εμείς συζητάμε να γίνουν κάποιες αλλαγέ στο κείμενο του Συμβουλίου για να ευθυγραμμίσουμε το κείμενο με τις θέσεις μας. Είναι πολύ πιο αδύναμη από την πρώτη ενάγνωση του Κοινοβουλίου, η οποία υποστηρίχθηκε τον Απρίλιο του 2009 με μια μεγάλη πλειοψηφία. Η θέση επίση τη Κομισιόν δεν δίνει καμία σαφήνεια αναφορικά με την νομική ευθύνη των ε, υλοτόμων και, των, ε, και όσων διαθέτουν ξυλία στην αγορά. και περιορίζει το θέμα του ορισμού. Δεν διευκρινίζει διάφορες ποινές ε, ή κυρώσεις ε, για, σε επίδοση παραβάσεις ε, και προβλέπει ένα ε, μείγμα, ένα μεικτό καθεστώς, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο χαλαρό αυτό που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Για να ενισχύσουμε λοιπόν τον κανονισμό και να πετύχουμε τους στόχους για την πρόληψη της εμπορίας παράνομα λειτουργημένης ξυλίας και πρωινού εγώ έχω αναδιατυπώσει πολλά από τα στοιχεία στην πρώην του στο Κοινοβουλίο. Να σας συνοψίσω τις βασικές ιδέες Κλείνω ανάμεσα στι θέσεις ε, του Συμβουλίου και των προτάσεων μου. Η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ περιοριστική και δεν πάει ιδιαίτερα μακριά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η θέση του Συμβουλίου επικεντρώνεται σε ένα και μοναδικό σημείο σε ό,τι φορά την ε, εμπορία ξυλίας. Μόνο όσοι ε, παρέχουν, ε, ούτε μπορούν παράνομα λειτουργημένη ξυλία ε, πρέπει να εφαρμόσουν το σύστημα της σε επιμέλεια, τη υποχρεωτικής επιμέλεια. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις σχετικά με το θέμα της νομιμότητας αυτών των προϊόντων ξυλίας. Επίσης δεν απαγορεύει την εμπορία παράνομη λειτουργημένα ξυλίας και ε, εισάγει την έννοια του αμεληταίου κινδύνου και ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ε, ικανοποιεί διόλου. Αυτό είναι κάτι επίσης που είχαμε εξετάσει το 2003. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η θέση του Συμβουλίου ως έχει θα μπορέσει να πετύχει τον στόχο μας και να διασφαλίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αγορά σχετικά με την ξυλία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να εκδώσουμε μια συγκεκριμένη ρητή θέση που θα αφορά την απαγόρευση της εμπορίας ε, παράνομα αλυτωμένης ξυλίας και πρώην ξυλίας, ε, όπως έχουμε εξάλλου προτείνει. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στο Lacey Act των Ηνωμένων Πολιτειών του που ε, ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια, το Μάιο 2008. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την δέουσα επιμέλεια, την... ειδικά σε ό,τι αφορά τους, τα άτομα που διαθέτουν στην αγορά ξυλία και προϊόντα ξυλίας για πρώτη φορά, θα πρέπει λοιπόν να φέρουν την ε, μέγιστη ευθύνη. Επίση ε, κρίνω ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε τα όσα είχαμε συμπεριλάβει στην πρώτη μας ανάγνωση, δηλαδή να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ε, φορέων που διαθέτουν στην αγορά ξυλία και προϊόντα ξυλία, δηλαδή καθιστούν διαθέσιμε στην αγορά για πρώτη φορά και αυτού που διαθέτουν στην αγορά ε, προϊόντα ξυλία. Αυτή η διάκριση λοιπόν μας οδηγεί στο ότι μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικές απαιτήσει από του φορείς εγώ συμφωνώ με την θέση του Συμβουλίου ότι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά ξυλία και πρώτη για πρώτη φορά θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρω ε, την δέουσα επιμέλεια και αυτοί οι οποίοι διαθέτουν ε, τα προϊόντα ξυλίας ε, παρανόμως θα πρέπει να υπόκειται σε κυρώσεις και θα πρέπει λοιπόν και θα πρέπει λοιπόν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, εκδηλασιμότητα των ε, προϊόντων αυτών και νομίζω θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πολλοί ε, φορείς στην Ευρώπη έχουν ήδη αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες. Αυτή η υποχρεωτική επιμέλεια ε, χρησιμοποιείται και για ένα άλλο στόχο. Φροντίζει να ε, μειώσει, να μετριάσει τις ε, παραβιάσεις και τις παραβάσεις. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν αυτό το θέμα της δέουσας επιμέλειας σε όλη την σημασία που έχει για όλη την αλυσία, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Δανία ε, επιθυμούν να καλυφθούν από αυτό μόνο όσοι διαθέτουν στην αγορά ξυλία και προϊόντα ξυλία για πρώτη φορά. Το, σύμφωνα με την ε, θέση του Συμβουλίου, το υπόθεση δεν πάει και πολύ μακριά. Αναφέρεται μόνο ο πρώτος ε, φορέας ε, που διαθέτει αυτά τα προϊόντα. Και επίσης δεν ε, επιτρέπει την χνηλασιμότητα την οποία εμείς επιθυμούμε. Δηλαδή το παράνομη υλοτομημένη ξυλία μπορεί να διατίθεται στην αγορά χωρίς ε, να επιβάλλονται κυρώσεις. Κάθε λοιπόν ε, παρανομία θα πρέπει να υπόκειται σε κυρώσεις και πρόστιμο. Αντί λοιπόν να αναφερθούμε στον πρώτο φορέα, θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη απαγόρευση σύμφωνα με την επέκταση της, ε, επέκταση της διεύθυνσης επιμέλειας. Και είναι αυτό το οποίο προτείνω. Κάτι ακόμα προτού να ολοκληρώσω. Να τονίσω ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα σε ό,τι αφορά την δέουσα επιμέλεια και την προσέγγιση την απαγορευτική. Συνδυαζόμενα καλύπτουν το κενό που υπάρχουν και αυτός ο συνδυασμός ασκεί άλλη πίεση και οι φορείς θα, θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την δέουσα επιμέλεια σε όλα τα επίπεδα το γεγονό ότι κάθε φορέα θα μπορέσει να διωχθεί για την παράνομη λοτομία αυτό θα ε, οδηγήσει στο να, έχουμε, να παρέχονται στις αγορές μας ε, μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλία. Και η νομοθεσία θα μπορεί να εφαρμόζεται πιστά. Η δέουσα επιμέλεια υφίσταται ήδη όπως στην, με ένα παράδειγμα στην οδηγία περί ξεπλήματος των χρημάτων. Τώρα, επανερχόμενοι στην, στην νομοθεσία που εφαρμόζεται, να πούμε ότι το σχέδιο δράση FLEGT δηλώνει ότι ο ευρύτερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ενθαρρυνθεί η αηφόρο διαχείριση των δασών και δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη παράνομη υλοτομία με ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό ο κανονισμό, ο FLEGT, θα μπορέσει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τι διατάξει που έχουν υπογραφεί και σε διεθνέ επίπεδο για να συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο τη αηφόρων ανάπτυξη ω μέσο αντιμετώπιση των αιτίων τη παράνομη υλοτομία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε ό,τι φορά τον ορισμό της, της ε, νομοθεσίας θα ήθελα να στηριχθούμε στο σχέδιο δράσης FLECT αλλά και στην προσέγγιση Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, VPA. Πολλές χώρες ε, διαπραγματεύονται ή διαπραγματεύτηκαν το σχέδιο δράσης ε, FLEGT με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε λοιπόν να ε, ζητήσουμε και από άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο δράσης να συμμετάσχουν με βάση τις ε, εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης VPA. Αφετέρου, έχοντας έναν στόχο που είναι τόσο ευρύς όσο και αυτός ο οποίος προβλέπεται στο σχέδιο δράσης ε, FLEGT και VPA, θα ζητήσω ότι θα πρέπει να ε, προωθήσουμε αυτές τις συμφωνίες Και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δοθούν κατευθύνσεις γραμμές στα κράτη-μέλη ώστε να δείξουν ε, αυστηρότητα στην εφαρμογή αυτών των ποινών. Θα πρέπει να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές ε, οι κυρώσεις αυτές, να είναι ιδιαίτερα αυστηρές έτσι ώστε να μην υπάρξουν κάποιες ε, σημεία αδυναμίας Γι' αυτό επανεισάγω τα βασικά στοιχεία που περιείχαν στην νέα, πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου όπως ε, και ζητάω να εφαρμοστούν οι ίδιες κυρώσεις που εφαρμόζονται στην παράνομη και λαθρέα αλία. Για να υπάρξουν εναρμονισμένα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της ε, παρακολούθησης του συστήματος της δέουσας ευμέλειας θα πρέπει να εφαρμόζονται και να γίνονται οι έλεγχοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενιαία και διάφανη εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Και τέλος, το Συμβούλιο εισάγει δύο εξαιρέσει για τα ανακυκλωμένα προϊόντα και για το λεγόμενο αμεληταίο κίνδυνο. Τώρα, σε ό,τι φορά τα εγκυκλωμένα προϊόντα, δεν είναι διόλου σαφέ όπω είναι διατυπωμένο το κείμενο τώρα, τι, εννοούν, τι εννοεί το Συμβούλιο με τα ανακυκλωμένα προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ παραμένω ανοιχτή σε συστάσει που θα ανεφέρονται ότι τα ανακυκλωμένα προϊόντα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, αλλά η διατύπωση θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάσει την ακαιρεότητα της νομοθεσίας. Εγώ προσωπικά ζήτησα να διαγραφεί διότι θεωρώ ότι ε, αποτελεί μια κερκόπορτα στην νομοθεσία. Αν δεν υπάρχει ένα σαφή ε, ε, αυτή η έννοια των αντικλωμένων προϊόντων και της εξαίρεση τους θα επηρεάσει το σύστημα της δέουσα επιμέλεια. Τέλος, το θέμα της του ελέγχου και της πιστοποίηση. Γνωρίζω ότι πολλέ οργανώσει έχουν ε, τονίσει ότι θα πρέπει να ε, κάποιες εξαιρέσεις ε, από την πιστοποίηση. Αλλά θεωρώ ότι μια γενική εξαίρεση θα ήταν ανεπαρκέστατη, διότι δεν θα ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο θα εξαιρείται σε ό,τι φορά την πιστοποίηση εάν θα έχουν τα προϊόντα αυτά πιστοποιητικό ή σίτες. Να πούμε ότι τα προϊόντα ξυλίας που μπαίνουν στην αγορά με πρότυπα φλέκ ή σίτες ε, μπορούν να αποτελέσουν εξαίρεση σύμφωνα με τον κανονισμό, αλλά αυτό δεν αφορά όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα. Λοιπόν, εάν υπάρξει μια γενική εξαίρεση, αυτό σημαίνει ότι θα αποκλειστούν όλα τα προϊόντα από οποιοδήποτε έλεγχο. Ακόμα και αν οι αρμόδιες αρχές εντοπίσουν παράνομη υλοτομία σε κάποια περιοχή, δεν θα μπορεί να αναλυφθεί νομική δράση κατά αυτών των εταιριών ή των ατόμων που διαθέτουν τα προϊόντα και μια απόλυτη εξαίρεση δεν θα ήταν η κατάλληλη λύση. Καταλήγοντας πιστεύω ότι η θέση του Συμβουλίου δεν είναι αρκετά αυστηρή για να ε, την να αποτρέψει την ε, εμπορία παράνομης, παράνομα υλοτομημένα ξυλίας. Νομίζω ότι οι συστάσεις μου είναι καταλληλότερες και παρακαλώ να τις δεχτείτε και αν τις εγκρίνετε. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για την εξαντλητική παρουσίαση ενός ε, ιδιαίτερα σημαντικού θέματος. Νομίζω πως εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την θέση σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους. Αν μπορείτε λοιπόν να παραμείνετε εντός ενός τριλέπτου ο καθένας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινάμε από τον κύριο Ασθένη. Ε, It's a legislation that... Πρόκειται για μια νομοθεσία που πραγματεύεται τις υποχρεώσεις για τους παρόχους στον ε, τομέα της αγοράς της ξυλίας. Αλλά φυσικά όλα έχουμε κατά νου την αλλαγή του κλίματος και κοιτώντα και λαμβάνοντα υπόψη την αποτυχία της συνόδου της Κοπενχάγης φαίνεται ότι θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αλλά και ο καθένας ε, στην εθνική του επικράτητα. Και τμήμα αυτής της δουλειάς είναι να σταματήσει η εισαγωγή παράνομης υλοτομίας, να σταματήσει η αποψήλωση, η οποία ευθύνεται για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών. Και έχουμε χώρες όπως η Βραζιλία, η οποία είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο, στη ρήπανση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι το 30% της ηλεκτρομίας στην Βραζιλία και στην ε, Ινδονησία είναι παράνομη και στη Χιλή. Άλλες ε, αναλύσεις μιλούν για 80%. Στο Κονγκό έχουμε πιο πολλές εκπομπές από ότι το Βέλγιο, η Ελλάδα και ούτω καθεξής και πολλές άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση λοιπόν της αποψήλωσης αποτελεί ένα τρόπο άμεσης αντιμετώπισης της μείωσης της εκπομπής ε, αερίων του θερμοκηπίου. Όπως είπε η Καρολάιν, το Συμβούλιο αγνόησε την πρώτη μας ανάγνωση από τις 88 τροπολογίες, 98 τροπολογίες μόνο, δύο πέρασαν, δύο από τις 98, τονίζω. Και αυτό βελτίωσε κατά κάποιο τρόπο τον ορισμό της νομιμότητας στην πρόταση του Συμβουλίου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον αμελταίο κίνδυνο, τον οποίο θεωρώ ως μια τεράστια παγίδα. Και επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν ε, η έλλειψη της απαγόρευσης και πολλά άλλα προβλήματα. Φαίνεται ότι επικρατεί ο φόβος ότι η απαγόρευση θα συνεπαγόταν τεράστιο κόστος για τις εκάστοτε κυβερνήσεις μας. Και ζήτησα σχετικέ εκτιμήσεις. Καμία χώρα δεν έχει τέτοιες εκτιμήσεις. Η ευρωπαϊκή εκτίμηση είναι σαφής. 116 εκατομμύρια ευρώ για τα 27 κράτη-μέλη. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το ποσό αυτό με την εκτίμηση του τι πληρώνουμε για να αντιμετωπίσουμε την αποψήλωση με χρήματα το Fast Track, 2 δις ευρώ, πραγματικά είναι αμεληταίο το ποσό. Κλείνω λέγοντας το εξής. Δύο θέματα θα ήθελα να τονίσω για, τα, για την πρόταση της Καρολάιν, η οποία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να είναι καλύτερος όμως ο σύνδεσμος, αν θέλετε, η σύνδεση μεταξύ της απαγόρευσης και του συστήματος της δέουσας επιμέλειας. Γιατί έτσι θα διασφαλιστεί η απαγόρευση μέσω της δέωσης επιμέλειας. Αυτό θα πρέπει να εκφραστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και επίσης να κινηθούμε πιο πολύ προς ε, την νομοθεσία FLECT. Να υπάρχει μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα. Το FLECT ε, είναι ένα μέσο το οποίο ε, λειτουργήσε και συμπεριλαμβάνει την ε, συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών έχει σχετική τεχνογνωσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η εμπειρία. Merci. Ε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 ξεκίνησε με τις προτάσεις για τον κανονισμό αυτό, έγραψε ότι η παράνομη ηλεκτριμία εξακολουθούσε να αυξάνεται και σε κάποιες χώρες η ποσότητα της παράνομης ξυλίας είναι πιο υψηλή από ότι αυτή της ε, νόμιμης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε είτε συμπέρανε ότι θα έπρεπε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Πριν ε, από δύο εβδομάδες η ΦΑΟ εξέδωσε μία νέα σύσταση και μία νέα ανάλυση για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο και παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί κατά κάποιο βαθμό η υλοτομία, η ΦΑΟ θεωρεί, εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι ανησυχητικά υψηλά τα ποσοστά της παράνομης υλοτομίας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαπίστωση της ε, πρώτης πρότασης συμπέρανε ότι θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ μιας απαγόρευσης ή ενός συστήματος ε, ε, δέουσας επιμέλειας, due diligence. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε επέλεξε το σύστημα της δέουσας επιμέλειας, όχι αυτό της απαγόρευσης. Όπως ε, είπε και η συγγύτρια η κυρία Λούκας, μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο συστήματα χωρίς πρόβλημα. Αυτό της απαγόρευσης και αυτό της δέουσας επιμέλειας. Και όπως είπε και η συγγήτρια, σε πολλούς τομείς εφαρμόζεται το σύστημα αυτό στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα δύο συστήματα αυτά δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Εγώ θεωρώ και είμαι πεπισμένος ότι όλη η κοινωνία κινείται προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και ότι οι απαιτήσει ω προ την δέουσα επιμέλεια δεν χρειάζεται ε, να ορίζονται νομικά. Εφαρμόζονται ήδη από την αγορά και το βλέπουμε αυτό και από τους μεγάλους ε, φορείς οι οποίοι λένε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το σύστημα δέουσας επιμέλεια γιατί εφαρμόζουν ήδη τους σχετικούς κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν και προβλήματα και θα ήθελα να θέσω το θέμα των ε, του διοικητικού άχθους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μας πούνε οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό για τις μικρές επιχειρήσεις. Μπορούν πλέον να πληρούν όλες τις διοικητικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα συστήματα τα οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ή μήπως οι μικρές εταιρείε εισαγωγής ξυλίας δυσκολεύονται υπερβολικά. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί εύρυθμα, αλλά θα περιορίσει και στο ελάχιστο το διοικητικό άχθος. Τέλος, Πρόεδρο, θεωρώ ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε μια στεναρή γραμμή, γιατί όπως είπα εξ αρχής, το πρόβλημα είναι τεράστιο, το πρόβλημα της αποψήλωση. Και δεν μιλάμε μόνο για τα δάση, μιλάμε και για το κλίμα, όπως είπε και ο συνάδελφο Αρσένης. Μιλάμε όμως και για το θέμα της ε, ελάττωση τη βιοπικιλότητας. Λοιπόν, στο δύο αυτό, στα δύο αυτά θέματα... Φυσικά όλα τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την ίδια γραμμή. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υποβάλλει τόσο αδύναμη πρόταση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην κοινή θέση. Το καλό είναι ότι ακούμε καλές ειδήσει ε, ότι στο Συμβούλιο εκφράζονται ανησυχίες και ότι πολλές ε, χώρες θα ήταν υπέρ μιας απαγόρευσης. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε ένα μικρό σπρόξιμο, αν θέλετε, ως Κοινοβούλιο για να κινηθεί το Συμβούλιο προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την εισηγήτρια για αυτήν την ε, νομοδότηση, στην οποία με η εισηγήτρια. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, αφού δεν συμμετείχα στο τελευταίο κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για ένα σύστημα με την εφαρμογή της εδέουσας επιμέλειας, με αυτό το due care, και νομίζω πως ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια μακρά ιστορία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία συμπαγών, αν θέλετε, νομοθετικών προτάσεων. Δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε εδώ κάθε κενό και νομίζω πως η συγκήτρια έκανε εδώ μια πολύ καλή δουλειά για να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Ε, εγώ ανησυχούσα πολύ και νομίζω πως όλοι όσοι έχουν αναμειχθεί σε αυτή τη διαδικασία ανησυχούσαν γι' αυτό, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή πώς οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να τηρήσουν όλους αυτούς τους κανόνες που αποβλέπονται από την νομοθεσία χωρίς να προκύψει επιπρόσθετο κόστος. Και άκουσα ανησυχίε από πολλές επιχειρήσεις ότι υπάρχουν αυτέ οι ανησυχίε για αυξημένο κόστο, αλλά όταν ε, ζήτησα περισσότερε εξηγήσει να μα πούνε δηλαδή ποιο είναι αυτό το επιπρόσθετο κόστο, υπήρχε απόλυτη ησυχία. Δεν έλαβα απαντήσει, γιατί δεν βλέπουμε. Δεν είναι σαφέ το ποιε ακριβώ θα είναι οι περαιτέρω εργασίε που θα χρειαστούν οι οποίε θα επιφέρουν αυτό το κόστο. Άρα λοιπόν η δημιουργία ενό τέτοιου συμπαγού συστήματο δεν νομίζω πω είναι επιφέρεια υποχρεωτικά και επιπρόσθετο κόστο. Και σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, τις ε, καλύτερες ποιότητες πληροφορίες οι οποίες θα διαβιβάζονται εφαρμόζοντας σε μάκρο επίπεδο την ε, δέουσα επιμέλεια είναι κάτι το οποίο νομίζω πως θα συμβεί με έναν τρόπο πολύ ομαλό. Νομίζω πως οι τροπολογίες που έχουν πρόταθει από την εισηγητριά μα είναι οι σωστέ, δηλαδή θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, δεν είμαι εγώ σκιώδης από την πλευρά του ΕΛΚΑ, επειδή, επειδή ο συνάδελφος ο αρμόδιος ο κ. Ε, θα ήθελα να πω εδώ ε, κάποια πράγματα. Ε, κύριε Λουκασά, έχετε εδώ την δική μας ε, υποστήριξη. Ε, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε ο συνάδελφο από του φιλελεύθερου σε ό,τι αφορά τι προσπάθειέ μα για να μειώσουμε και μάλιστα πολύ δραστικά την παράνομη λοτομία. Εδώ πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα. Ε, το ζητούμενο εδώ είναι το κατά πόσο αυτά τα όσα προτείνατε εσεί με τόση μεγάλη προσοχή πράγματι θα οδηγήσουν σε μειωμένε εισαγωγέ παράνομα λοτομημένη εξηλία. Ε, και εγώ πραγματικά εδώ βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ νομίζω δηλαδή πως εδώ το βασικό σημείο είναι η συνείδηση, αν θέλετε, η, ε, το σκεπτικό, αν θέλετε, των κρατών μελών να μην επιθυμούν δηλαδή να εισάγουν την ε, παράνομα ελωτομημένη ξυλία. Και μόλις τώρα το ακούσαμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτό, είναι οι αρμόδιες κρατικές αρχές οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει αυτή τη συνείδηση, δηλαδή του σωστού, του δέοντος ελέγχου τη εισαγόμενη ξυλία. Και επειδή ακριβώ αυτέ οι αρμόδιε κρατικέ αρχέ δεν προβαίνουν στου απαραίτητου ελέγχου, προσπαθούμε εμεί να πάμε εδώ σε ένα σύστημα, αν θέλετε, ετικετοθεσία ή τι θέλετε, πώ θέλετε να το πω, εν πάση σε μια γραφειοκρατική διαδικασία όπου χρειαζόμαστε περισσότερα έγγραφα. Για να δούμε όμω τι θα συμβεί τελικά σε ένα σημείο λεωτόμηση, δηλαδή πραγματικά εκεί. Τι να βάζουμε, να βάζουμε ένα σήμα, αν θέλετε, σε κάποιου κορμού δέντρων καλώ. Αλλά τι θα κάνετε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το πριονίδι, σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά επιμέρου, α λέτε, κομμάτια ξύλου. Δηλαδή εκεί τι, τι ακριβώ, τι, περιμένετε ότι θα μπει, πώ θα μπει εκεί το σήμα. Δηλαδή ε, α τα σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλα δηλαδή την ε, θετικά εννοούμενη βούλη στην οποία διακρίνω. Αντιλαμβάνομαι ότι πρώτη για μια πρόκληση εδώ για τα δάση και ούτω καθεξής. Αλλά πραγματικά ακόμα κι αν ε, πούμε ότι θα εφαρμόσουμε ένα ε, σύστημα που θα βάζουμε σήματα και ούτω καθεξής θα πρέπει ε, να δούμε να υπάρχει και ένας τρόπος επαλήθευσης, αξιολόγησης δηλαδή αυτού του συστήματος ετικετοθεσίας. Αλλά από εκεί μετά σας λέω υπάρχουν κομμάτια προϊόντα δηλαδή ξυλία τα οποία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε επιπρόσθετες υποχρεώσεις και εδώ θα πρέπει πάλι να τσακωθούμε, αν θέλετε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η δική τη αρμοδιότητα, να αναλάβει σωστά τι δικέ τη αρμοδιότητε. Δηλαδή να μην ε, ξεκινάει εδώ με περίπλοκου υπολογισμού. Όχι, εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει το τι συμβαίνει στα ίδια τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν δηλαδή εδώ τομεί όπου δεν συμβαίνει πραγματικά τίποτα από την πλευρά των κρατών ε, Και ναι, πράγματι ακούστηκε και από τον συνάδελφο ότι δηλαδή είχαμε το τροπολογίε, τώρα μόνο δύο ε, έγιναν ε, δεκτέ. Ε, τι, ποιο είναι το συμπεράσμα, δηλαδή ότι είναι χαζό το συμβούλιο και είμαστε εμεί οι έξυπνοι. Όχι, δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, Σα λέω, υπάρχουν όλα αυτά τα προϊόντα ξυλία, υπάρχουν οι ίδιε εφημερίδε, αν θέλετε. Πώ θα βάλουμε εκεί ένα σήμα προέλευση, αν θέλετε. Τι, να τι θα γίνει εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε ενδεχομένω σε μια μπριζόλα, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα Ατλαντικό, αλλά μιλάμε εκεί ε, για ένα διαφορετικό τομέα. Το στόχο μα πάντω θα πρέπει να είναι κοινό, δηλαδή καλύτερο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών και προφανώ η αρχή τη δεούσα επιμέλεια εδώ έχει νόημα. Ασχύει όμω κυρίω για τι τελωνιακέ αρχέ. Κατά συνέπεια ισχύει για τι δικέ μα εθνικέ κυβερνήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φλόρεν. Ο Chris Ντέιβι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν, μιλούσε, αν μιλούσαν όλοι οι Βρετανοί συντηρητικοί με το ίδιο πνεύμα που μίλησε και η συνάδελφο, δεν θα ανησυχούσα για το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών που ανακοινώθηκαν σήμερα στην Βρετανία. Δυστυχώ ξέρουμε ότι μάλλον υποεκπροσωπείται το είδο τη Τζούλη στη Βρετανία ευχαριστώ πάντως, ε, την ευχαριστώ για ε, τα σχόλιά της, την ευχαριστήσω και την Καρλάν Λούκας. Είναι καινούργιο το κοινοβούλιο, αλλά το ίδιο θέμα το συζητάμε ε, πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε και στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα κοιτάξαμε τις προτάσεις FLECT και πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια δική της ατζέντα το θέμα και πολλοί ήταν αντίθετοι. Πολλοί στην Επιτροπή ε, υποστήριζαν ότι δεν θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε νομικούς περιορισμούς, αλλά νομίζω ότι πολλά από τα εμπόδια πλέον έχουν καταρρευθεί και είναι πιο ελεύθερη η σκέψη για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι διχασμένο από πολλές απόψεις για πολλά θέματα, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πολλοί, πολλοί κόσμος έχει την αίσθηση ότι είναι απλά λάθος να επιτρέπουμε εισαγωγές παράνομης υλοτομία που ξέρουμε ότι προέρχεται από παράνομες πηγές. Και οι καταναλωτές μας ε, αποτελούν, έχουν την αίσθηση ότι αυτό ε, μειώνει την βιοπικιλότητα, αυτό προκαλεί την παράνομη ηλεκτρονία. Οι προτάσεις FLECT είναι καλές μεν, αλλά πολύ αργές και πολύ απλά δεν καλύπτουν αρκετή, αρκετό από τον κόσμο, αν θέλετε, από την συνολική επικράτεια που μας απασχολεί. Και είναι προφανές ότι πολλά σημεία επί του περιεχομένου θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική πολιτική, αν θέλετε, κατεύθυνση, μέσω του Κοινοβουλίου, μέσω της πρώτης ανάγνωσης, μέσω της εισηγήτριάς μας, έχουμε θέσει πολλές τροπολογίες για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο, διχασμένο μεν, αντιστέκεται. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ όλων των ομάδων για να προωθήσουμε το θέμα. Και καταλαβαίνω φυσικά ότι θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί, γιατί πολλά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αν δεν καταλήξουμε σε μια θέση όπου θα μπορέσουμε να ασκήσουμε πλήρως τα δικαιώματα στη συναπόφαση, ε, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ απογοητευτικό. Ας το προωθήσουμε λοιπόν και δείξουμε κάποια φιλοδοξία σε τελική ανάλυση. Peter Van Delen, si Παρακαλώ, αν μπορείτε να περιορίσετε κάποιες παρεμβάσεις σας και τη διάρκεια τους, γιατί είναι πολύ φορτωμένο σήμερα το απόγευμα μας και δεν θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Ευτυχώς ε, η συνάδελφος Γκίλεν δεν είναι μόνη της, γιατί στο στην ομάδα της. Πρέπει να πω ότι μας βρίσκει σε ότι αφορά το καλύτερο περιβάλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να υποστηρίξω και την κυρία Λούκας για την πολύ καλή της έκθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παράνομη υλοτομία έχει καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη και σε ό,τι αφορά τα οικοσυστήματα, τη βιοπικιλότητα που πλήττονται έντονα. Αλλά υπάρχει και μια οικονομική πτυχή που υπονομεύει τις επιχειρήσεις αυτές. Πρόεδρε, λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ως Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση υποστηρίξαμε μια στεναρία θέση. Δυστυχώς το Συμβούλιο, ωστόσο, δεν ε, και δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη θέση αυτή και θεωρώ ότι αποτελεί πρόκληση για μας να παραμείνουμε στεναροί έναντι του Συμβουλίου, να φροντίσουμε ότι και στο εσωτερικό του Συμβουλίου θα υπάρξει διαφορετική τοποθέτηση από διάφορες χώρες. Αυτό είναι κρίσιμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στο θέμα της απαγόρευσης σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές και την πώληση παράνομης ξυλίας και είδαμε και ότι υπήρξαν αποτελέσματα και στην Αμερική. Ας κινηθούμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή, ας υποστηρίξουμε μία αδιάλακτη θέση προκειμένου να τερματιστεί διαπαντός η παράνομη ξυλία και να μιλήσουμε με μία φωνή ως κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, ο Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά την προετοιμασία του θέματος αυτής, διάβασα πολλά έγγραφα περιβαλλοντικών ενώσεων, των κρατών μελών και από διάφορες άλλες ενώσεις και θα πρέπει να πω ότι όσο πιο πολλά διαβάζω, τόσο πιο πολύ ενοχλούμε και θυμώνω, γιατί και από τις δύο πλευρές ε, θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται και θεωρείται με πολύ μονόπλευρο τρόπο, γιατί στις περιβαλλοντικές ενώσεις βλέπω ότι λείπει η διάσταση του μικρού ιδιοκτήτη, των μικρών εκμεταλλεύσεων και σας μιλώ με την ε, εμπειρία που έχω από τη δική μου περιφέρεια, από την ε, Βορειοελληνία Βεσφαλία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εμπορία πολλών τέτοιων προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα για τη σωστή ε, διαχείριση των πόρων στους μικρούς εκμεταλλευτές. Δεν θα πρέπει να καταντήσουμε αντιπαραγωγική. Και σε πολλούς τομείς στην Ευρώπη, σε πολλές περιφέρειες χρειαζόμαστε πιο πολύ ηλετόμηση για να καταστεί το σύστημα ε, βιώσιμο. Από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά, η οικονομική πλευρά, μιλάει μόνο για τους μικρούς ε, αυτούς ε, φορείς. Μιλούν μόνο για το γραφειοκριτικό άχθος, δεν θίγουν όμως το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορώ και οι δύο πλευρέ δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στο σύνολό του. Φυσικά ισχύουν αυτά που είπε και η Καρολάιν Λούκα και ο Κρήτονας Αρσένη. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την παράνομη λετομία και είναι τεράστια η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν ανταποκρίνεται ω τώρα. Από την άλλη, θα πρέπει να ακούσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να διαπιστώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές αυτές τις καταστάσεις προκειμένου να βρεθεί μια εύλογη λύση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη λετομία και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πολύ πιο έντονα από ό,τι, από ό,τι τώρα. Και παράλληλα να προσέξουμε να μην επιβαρύνουμε χωρίς λόγο αυτούς που ω τώρα λειτουργούσαν στην αγορά χωρί πρόβλημα. Όλα αυτά σε ό,τι αφορά τι κυρώσει που ανέφερε η Καρβάνη Λούκα και εγώ είμαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής ρύθμιση, αλλά παράλληλα χρειαζόμαστε και μια ελάφρυνση, μια ευελεξία για τις μικρές επιχειρήσεις, όπου δεν υπάρχει πόνοια παράνομης υλοτομίας. Κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν συμμετείχα στις εργασίες του προηγούμενου Κοινοβουλίου, κατά το οποίο είχε συζητηθεί ε, παρούσα νομοθετική πρόταση, αλλά υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία σκέφτομαι. Προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από κάποιον άλλον και εμείς μπορούμε να αποτελέσουμε ένα μέρος αν θέλετε της λύσης αλλά όχι τη συνολική λύση. Είναι λοιπόν λαθασμένη προσέγγιση να προσπαθούμε να αποτελέσουμε τη μοναδική λύση όταν αποτελούμε μόνο ένα τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Φοβούμε λοιπόν ότι προσπαθούμε εδώ να επιτύχουμε μια συνολική 100% λύση όταν εδώ το πρόβλημα εάν θέλετε επιλύεται με μια αναλογία 80% προς 20%. Δηλαδή 80% του προβλήματος μπορεί να επιληθεί αν θέλετε με το 20% του συνολικού απαραίτητου κόστους και το, 20% και το υπόλοιπο μπορεί να επιληθεί και από τους υπολείπους που είναι υπεύθυνοι. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να γίνει να ληφθούν και μέτρα τα οποία βρίσκονται πιο πριν μέσα στην αλυσίδα της προμήθειας. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή πώς θα είναι σε θέση εκμεταλλεύσεις να τηρήσουν τέτοιες διατάξεις εάν δεν υπάρχει επιπρόσθετο κόστος. Αλλά δεν έχουν, αν θέλετε, την υποχρέωση για να ε, αποδείξουν ότι πράγματι υπάρχει αυτό το κόστο. Εμεί θα είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να πείσουμε τι επιχειρήσει ότι έχει νόημα να υπάρχει περισσότερο κόστο στο πλαίσιο αυτή τη νέα ε, νομοθεσία. Όχι σε ό,τι αφορά την αρχική διάθεση αυτών των προϊόντων στην αγορά, αλλά σε ό,τι αφορά ειδικότερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει οι οποίε εμπορεύονται ξυλία, δηλαδή αγοράζουν ξυλία από μια άλλη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτέ λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα πρέπει να έχουν με ελάχιστη αν θέλετε αξιοπιστία και αυτή η αξιοπιστία, αυτό το πλαίσιο αξιοπιστίας θα πρέπει να διασφαλιστεί, να παρασχεθεί από τι κυβερνήσει και από την κατάλληλη εφαρμογή τη παρούσα νομοθεσία. Δηλαδή, εάν δεν μπορούμε εμεί να σταματήσουμε την παράνομη λοτομία, ή μάλλον την παράνομα, παράνομα ενοοτοβημένη ξυλία από το να εισέλθει μέσα στη δική μας αγορά, γιατί να προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να επιβάλλουμε απαγορεύσεις ή να σταματήσουμε την προμηθευτική αλυσίδα στη μικρομεσαία επιχείρηση η οποία νομίμως έχει προμηθευτεί αυτή την ξυλία από μια άλλη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την διαπραγματευτική θέση την οποία θα πρέπει να λάβουμε στην Κοινοβούλιο, αλλά θα είναι ακόμα καλύτερη αν είμαστε λογικοί και αν η νομοθεσία που προτείνουμε είναι δίκαιη για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουμε ακόμα τέσσερις αγορητές. Παρακαλώ να παραμείνετε εντός ε, διλέπτου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα. Μαδαγασκάρη. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αναγνωρισμένη, ότι υπήρξε ένα πραξικόπημα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κονδύλια της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την παράνομη κυβέρνηση. Έχουν αρχίσει να αποψηλώνουν όλα τα πάρκα, όλους τους δρυμούς σου. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο ευθύνες. Πρώτα απ' όλα, οι εξαγωγής πρόκειται για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που μεταφέρουν αυτή την ξυλία και σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε, ατικές, σε ασιατικές. Λοιπόν, πώς να τιμωρηθούν εν λόγω έμποροι διότι συμμετέχουν στην παράνομη εμπορία αυτή τη ε, ξυλία. Και εδώ θα είναι ευθύνη και τα ευρωπαϊκά κράτη. Αν θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να επιβάλλουμε αποτρεπτικέ ε, οικονομικέ κυρώσει και στου εξαγωγεί και εδώ ερχόμαστε ε, αντιμέτωποι με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του και τα ευρωπαϊκά κράτη. Ευχαριστώ για την συντομία σας αλλά για τη σαφήνειά σας. Κυρία Γκρόστετ έχει λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα. Είναι σίγουρο πως ε, θα πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο στόχο για να καταπολεμήσουμε την παράνομη λιτόμηση των ε, δασών. Χρειάζεται λοιπόν μια υποχρέωση, μια υποχρέωση η οποία θα είναι ανάλογη με το επίπεδο του κινδύνου. Πρέπει να δείξουμε αποτελεσματικό και φαστικότητα για να καταπολεμήσουμε την παρανομία με την χορήγηση πιστοποιητικών τα οποία θα χορηγεί μια ανεξάρτητη πηγή. Και Χρειάζεται λοιπόν να αναφέρεται η προέλευση του ξυλίας. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω την έστασή μου στην τροπολογία υπερθούν 70 τη ηγέτρια που ζητάει τη συμπερίληψη των εκδοτών στον κανονισμό. Κυρία Λούκο ζητάει οι εκδότε να δείξουν λογική ε, ε, δέους επιμέλεια για τον θέμα της χρήσης ε, του ε, ξύλου το οποίο χρησιμοποιείται για τον χαρτοπολτό. Θα είναι δύσκολο στην περίπτωση αυτή να γίνει μια εξέταση αναλυτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν ως εκ τούτου να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την προέλευση, διότι ο χαρτοπολιτός που χρησιμοποιούν είναι χαρτοπολιτός που αγοράζει στις διεθνείς αγορές και οι προμήθειες συνεχώς εξελίσσονται και είναι δύσκολο λοιπόν να υπάρξει αυτή η χνηλεσιμότητα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Κάνει άποψή μου λοιπόν. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους εκδοτικούς οίκους και να επικεντρωθούμε στο σύστημα μιας λύσης η οποία θα ε, αφορά τις προσπάθειες που θα καταβάλουν οι φορείς και οι δημόσιες αρχές στον, σε αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στην ε, υλοτομία, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος πρώτος θέτει το προϊόντα στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν και εναρμονισμένοι έλεγχοι, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πρόεδρε για να είμαι σύντομη. Πρόεδρος, ευχαριστώ για την κατανόησή σας, αλλά σήμερα το απόγευμα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να εξετάσουμε. Κύριε Αγκροστέρη, μπορείτε να κλείσετε το μικροφωνό σας παρακαλώ, μην ακούγεστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν θα ήθελα να αναλυθώ ότι ο κύριος Λούκας είχε εδώ μια καλή πρόθεση, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε εδώ με την, την αγορά με την οποία έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή ε, μια μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και μιλάμε και για την προώθηση ε, μιας πρώτης ύλης η οποία είναι ανανεώσιμη, η οποία μπορεί ε, να μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν εδώ χρειαζόμαστε πρακτικές λύσεις. Ε, σε αυτές θα πρέπει να στοχεύσουμε και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε εδώ υπερβολική γραφειοκρατία. Θα πρέπει να δοθούν τα σωστά κίνητρα στα κράτη-μέλη, οι διατάξεις οι οποίες ισχύουν και τις οποίες προτείνουμε εδώ να, να εφαρμόζονται από την πλευρά τους και να υπάρχει σωστός έλεγχος στα σύνορα. Ένα συνολικός έλεγχος τώρα όλε τι αλυσίδε ε, προμηθεία, θα ε, δημιουργήσει δυσκολίε, θα έχει επιπρόσθετο κόστο και θα, δεν θα είναι εύκολη στην πρακτική εφαρμογή. Πράγμα το οποίο δεν θα έχει όφελο ούτε για τον ε, καταναλωτή, ούτε για τον κλάδο της εξηλίας. Ε, δηλαδή πραγματικά ε, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα υπήρχαν ε, αυξημένα μείον εκτήματα για την αγορά της εξηλίας συνολικά. Άρα λοιπόν αφού δεν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε πρώτον ελέγχους στα σύνορα των κρατών μελών, δεύτερον οι συναφεί διατάξει να εφαρμόζονται και θα πρέπει οι σχετικέ διατάξει να περιοριστούν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να συγχωνευτούν, ώστε να μην έχουμε, να μην, ε, αν θέλετε, παρεμβαίνουμε με τη δική μα νομοθεσία σε τρίτε χώρε. Ε, κάτι τέτοιο δεν νομίζω πω θα μα βοηθήσει. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει νόημα είναι να είμαστε ρεαλιστέ εδώ και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν και με το πρακτικό τρόπο τα όσα έχουν ήδη δεσμευτεί ότι θα τηρήσουν για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ε, σημαντική πρώτη την ξυλία γιατί νομίζω πως το θέλουμε όλοι αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένα είναι σαφές ότι κανένας δεν επιθυμεί την παράνομη ελοτομία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τροπικά δάση, αλλά το ζητούμενο είναι ε, ποια μέσα θα αξιοποιήσουμε για να το επιτύχουμε αυτό. Οι προτάσεις ε, της ε, εισηγήτριας τι σημαίνουν για την πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων και για τον σύνολο του κλάδου θα έλεγα μεγάλες επιβαρύνσεις που σημαίνει ότι δεν έχουμε επιπρόσθετη αξία από κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα δύο τρίτα της εισαγόμενης ξυλίας ή μάλλον της ξυλίας που εμπορεύονται είναι ε, χώρια πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, παρανομελοτόμηση. Άρα λοιπόν ε, με έναν τέτοιο τρόπο δεν είναι σίγουρο το κατά πόσο θα περιορίσουμε το ποσοστό της ε, παράνομα υλοτομημένης εξηλίας. Ε, δεν ε, αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί προτείνονται τέτοια μέτρα. Ίσως πέρα από την αρχή της δέουσας επιμέλειας να έχουμε να λαμβάνεται υπόψη ο, για παράδειγμα το είδος ε, του, της ε, ξυλίας, ε, η χώρα προέλευσης και ούτω καθεξής και να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης. Άρα λοιπόν ο αμεληταίος κίνδυνος και η σχετική αρχή θα μπορούσε να μα βοηθήσει να φτάσουμε μια, σε μια σωστή ισορροπία μεταξύ δηλαδή πρακτικών διατάξεων και μειωμένης γραφειοκρατίας. Ε, το να έχουμε ένα συνολικό έλεγχο είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο γραφειοκρατικό επίπεδο. Άρα λοιπόν η εισαγωγή από τρίτε χώρε με βάση την, ε, αν θέλετε, τη στάθμη τη επικοινωνία θα πρέπει να αξιολογούνται και νομίζω πω αυτό είναι ο τρόπος ε, για να προχωρήσουμε ώστε να φτάσουμε και σε ένα απτό αποτέλεσμα το οποίο ε, νομίζω πως θα ωφελήσει και τον ε, ευρωπαϊκό κλάδο της ξυλίας. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόσμπαχ, ε, λακωνικά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, μετά από τα όσα ακούστηκαν, να αναφερθώ στην παράνομη υλοτομία η οποία όμως ε, δεν φτάνει στην Ευρώπη, αλλά τη εκμετάλλευση εκμετάλλευσης επιτόπου και ενδεχόμενα να αποστέλλεται στην Κίνα. Εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε καμία δυνατότητα να εξακριβώσουμε ποιες είναι αυτές οι ποσότητες που εξάγονται προς την Κίνα, οι οποίες ε, αργότερα, σε μεταγενέστερο στάδιο, αποστέλλονται σε άλλα κράτη. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν έχουμε καμία ένδειξη και δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο. Αυτές οι ποσότητες ξέρουμε ότι μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Θα χρειάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τροπή να βρει τρόπους και μέσα για να συνάψει συμφωνίες συνεργασίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, εξάγουν και εισάγουν παράνομο λετωμένη ξυλία έτσι ώστε δεν θα είμαστε εμείς μόνοι μας οι οποίοι θα καταρτίζουμε κανόνες συγκεκριμένους οι οποίοι θα κοστίζουν και πολύ διότι σίγουρα έχουμε μια καλή πρόταση αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω ότι δεν ισχύει. Πρόεδρος, ε, τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν, κύριε Τζον Μπαζίλε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank um, Σας ευχαριστώ και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παράνομη υλοτομία και εργαζόμαστε εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά το σύστημα FLECT, σε ό,τι αφορά διμερείς συμφωνίες, αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω νομοθεσία. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να αναφερθώ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που μας τέθηκαν. Από τον κύριο Σεμπράντη, σε ό,τι αφορά το κόστος και τις συνέπειες ε, της ε, απαγόρευσης για τις μικρές επιχειρήσεις και κατά πόσο θα μπορούσαν να συνδυαστούν τα δύο συστήματα, τις δέωσες επιμέλειας και τις απαγόρευσης. Όπως ε, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το σύστημα της απαγόρευσης όπως ε, ονομάζεται, αλλά κατέληξε σε μια διαφορετική προσέγγιση, την προσέγγιση της δεύτερης επιμέλειας ε, από πλευράς των ε, φορέων εκμετάλλευσης. Για πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων ήταν να δοθεί μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στους φορείς, να γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν. Και για πρακτικούς λόγους γιατί το να αποδείξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά πόσο ένα κομμάτι ξύλο στην Ινδονησία κόπηκε, ε, υλοτομήθηκε παράνομα ή νόμιμα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στις μικρές επιχειρήσεις. Πολλά εξαρτώνται από το κατά πόσο η απαγόρευση αυτή θα συνδυαστεί με υποχρεώσεις για τους ε, φορείς εκμετάλλευσης στην υπόλοιπη αλυσίδα εμπορίας. Γιατί αν ο ε, εκμετάλλευσης μια επιχείρηση ε, διαθέτει άμεση επαφή με την πηγή, είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αν εμπλέκονται περισσότερες επιχειρήσεις, προφανώς αυτό θα πολλαπλασίαζε το διοικητικό άχθος για τα υπόλοιπα θέματα. Συμφωνούμε με την θέση της Καρλάιν Λούκας για την πιστοποίηση ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει γενική εξαίρεση για τα πιστοποιημένα προϊόντα. Και γενικά να έχουμε υπόψη μας προκειμένου νομοθεσία και οι απαιτήσει που θα από την κείμενη νομοθεσία να μπορούν να εφαρμοστούν από τους φορείς εκμετάλλευσης, να μην αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, υπερβολικά θεωρητικές ε, φιλοδοξίες. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το καθεστώς αναγνωρίση των ε, οργανισμών, δηλαδή εποπτείας, συμφωνήσαμε να λειτουργούν στα πλαίσια των κρατών μελών οι οργανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου και η πιστοποίηση που δίνουν λειτουργούν καλύτερα σε τοπικό επίπεδο, σε κράτος μέλος. Και παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι τέτοιοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να φέρουν κεντρική πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ζητήσω από την εισηγήτριά μας ε, να λάβει το λόγο προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ την, για μια ακόμα φορά για την υψηλή ποιότητα της εργασίας της. Κυρία Λούκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Μερικές ε, παρατηρήσεις. Πολλοί ανέφεραν ότι τον νόμιμα, νόμιμη ηλεκτρονημένη ξυλία είναι ένα καλό προϊόν. Εντίθετη ε, την περίπτωση δεν είναι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σχετικά με την παράνομη και νόμιμα ηλεκτρονημένη εξηλεία. Τώρα, αυτό δεν είναι θέμα που αφορά τι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει παράνομα ηλεκτρονημένη ξυλία. Τώρα, μερικά σχόλια σχετικά με τα όσα είπε η Κομισιόν πολλοί, συμπεριλαμβανομένοι και πέντε μελών του Συμβουλίου, συμφωνούν ότι η προσέγγιση της δεύτερης επιμέλειας από μόνη δεν θα μας εγγυθεί ότι δεν θα έχουμε παράνομη, παράνομη λειτουργημένη ξυλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει έλεγχος των φορών εκμετάλλευσης που διαθέτουν στην αγορά ξυλία και προϊόντα ξυλία. Ε, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η ω επιμέλεια δεν πρόκειται να πετύχει από μόνη τη τον στόχο. Η Κομισιόν αναφέρθηκε επίση και το πεδίο εφαρμογή ε, τη νομοθεσία. Α καθέσουμε σαφέ λοιπόν περί τίνο πρόκειται. Μιλάμε για την επιβολή νόμων οι οποίοι εφαρμόζονται στις χώρες όπου υλοτομείται η ξυλία. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε μια οδηγία σχετικά με το χρόνο εργασία στην Ινδονησία. Μιλάμε για την νομοθεσία που αυτή η τρίτη χώρα έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στην ε, επικράτειά της. Αυτό δεν είναι απίθανο να συμβεί και ένα από τα κλειδιά είναι ότι δεν ζητάμε για λιγότερο στο πλαίσιο του κανονισμού από ό,τι περιέχεται στις συμφωνίες Φλέκ. Διαφορετικά θα δημιουργήσουμε μια στρεβλή εικόνα και θα φροντίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη να περιορίσουν το εύρος της ε, τους νομοθεσιευτές τώρα. Θα σας ζητήσω να δείτε τι αναφέρεται ακριβώς στην έκθεση και όχι τι πιστεύετε πως αναφέρεται, διότι οι υποχρεώσεις που υπάρχουν είναι οι υποχρεώσεις της δέουσας επιμέλειας, η οποία δεν εφαρμόζεται σε όλους, αλλά μόνο σε όσους διαθέτουν προϊόντα στην... και προμηθεύουν την αγορά για πρώτη φορά. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζετε από πού προέρχεται το προϊόν σας και πού πωλείτε. Δεν είναι αυτό ιδιαίτερο άχθος, ούτε δημιουργεί περαιτέρω φόρτο εργασίας. Αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε σαφές ότι δεν είναι κάτι το δαπανηρό, είναι ένα απλό ζήτημα που ε, περισσότερες από τις επιχειρήσεις ήδη εφαρμόζουν. Έγινε ένα σεμινάριο σήμερα το μεσημέρι και είχαμε, είχαμε σε επαφή με τους με διάφορες οργανώσεις όπως το ΑΚΙΑ, το Καρφούρ κλπ. Και, και αυτή είναι υπέρ της δέουσας επιμέλειας. Το ότι έχουμε τώρα μια σειρά επιχειρήσεων που παίρνουν μια θέση πολύ πιο προοδευτική από αυτή του Συμβουλίου και της Κομισιόν, νομίζω ότι αποτελεί ένα μήνυμα. Αποστέλνουν ένα μήνυμα. Λοιπόν, αν αυτή η προσέγγιση για την οποία μιλάμε εδώ, ειδικά με την απαγόρευση είναι τόσο δαπανηρή. Πιστεύετε ότι οι ε, Ρεπουμπλικανοί θα τον είχαν ψηφίσει όταν ψηφίσανε πριν από δύο χρόνια τον νόμο στι στις ΗΠΑ. Ορισμένοι πρότειναν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τις ε, ζήτημα σε ό,τι φορά τις μικρές επιχειρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι υποχρεώσεις που τους ζητάμε είναι τόσο δαπανήρες δεύτερον. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες ιδέες όπως έχουμε το προηγούμενο με το REACH. Έχουμε κάποια help desk για να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις και ίσως και κάποια τεχνική ή οικονομική υποστήριξη θα τους βοηθούσε. Αυτό ίσως να απέτυχε και τέλος σχετικά με τη στρατηγική. ο Chris Davis είπε πολύ σωστά ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια στεναρή στέση εδώ στο Κοινοβούλιο αν θέλουμε να πετύχουμε το οτιδήποτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο έχουμε είχαμε μια πολύ ισχυρή θέση στην πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι αυτή τη θέση θα πρέπει να διατηρήσουμε. Φυσικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αλλά εάν πάμε με μια ε, πιο νερωμένη θα έλεγα θέση, δεν ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο. Λοιπόν, θα πρέπει να καταδείξουμε ότι δεν είναι δαπανηρό αυτή η νομοθεσία, δεν προκαλεί περαιτέρω άχθος, χρειάζεται υπάρχει δυνατότητα ε, χνηλασιμότητας, αν δεν υπάρχει τότε δεν θα πετύχουμε τον στόχο μας, χρειάζεται λοιπόν να διατηρήσουμε τη συνεργή μας θέση απέναντι στο Συμβούλιο. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Επενθυμίζω πω η καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση τροπολογιών είναι η 8 Απριλίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ε, ανάμεσα στι 26 και 28 Απριλίου και στην Ολομέλεια 17 ε, και 20, έως 20 Μαΐου. Ε, έκανα λάθος, δεν τα είπα σωστά. Συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα λάθος. Καταληκτική ημερομηνία, ναι, 8 Απριλίου, στην Επιτροπή 4 και 5, 3 και 4 Μαΐου και την Ολομέλεια θα περάσει τον Ιούλιο. Τώρα περνάμε στο επόμενο ζήτημα που αφορά την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια διαδικασία ιδιάζουσα διότι έχουμε ενστασία από πλευρά πρασίνων. Προτείνω λοιπόν, εάν συμφωνείτε για να διοργανώσουμε τις συζητήσεις μας, πως ενδεχόμενα ο Κλωτ Τέρμες να μας αναφέρει την ένσταση των πρασίνων ή οποιοδήποτε άλλος, η Κομισιόν να απαντήσει, να ξεκινήσει με τη συζήτηση αφού οι δύο υπόψη, ε, αφού ληφθούν υπόψη δύο θέσεις. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν στις 5 παραδέαρτο να έχουμε ολοκληρώσει το σημείο 5, διότι έχουμε άλλα δύο μεγάλα ζητήματα και το θέμα της αναφοράς αναφορικά με τη διάσκεψη της Ντόχα. Λοιπόν, ποιο ε, θέλει να εκφράσει την αίσθηση των Πρασίνων, Κλοντ Τιουρμέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. Για να καταλαβαίνετε άμεσα αυτά που λέω, κατευθείαν. Νομίζω ότι προκειμένου να κατανοήσουμε όλο το θέμα θα πρέπει να κοιτάξουμε τι συνέβη το 2008 όταν το σύστημα ETS ήταν υπό για την ε, αποθήκευση άνθρακα. Τότε εισήχθη η ιδέα να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθούν κονδύλια 300 εκατομμυρίων για να χρηματοδοτηθούν αφενός ε, η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα και κατά δεύτερο ε, μια σειρά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τότε όλες οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας βοήθησαν ουσιαστικά να περάσουμε τη συμφωνία αυτή. Τότε λοιπόν θεωρούσαμε ότι η αξία των 300 εκατομμυρίων θα ανερχόταν στα 7-8 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί θεωρούσαμε ότι η τιμή ανατόνων διεξιδίου του άνθρακα στο σύστημα ETS θα ήταν 25-30. Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, μεσολάβησε η οικονομική κρίση. Η βιομηχανία περνάει φάση ύφεση, χρειάζεται λοιπόν λιγότερα επιστοποιητικά, πέφτουν οι τιμές και έχουμε και το μπλοκ του την Ιταλία, δηλαδή την Πολωνία και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες ε, αντιστέκονται και έτσι και αυτό εμποδίζει την άνοδο των τιμών. Μία πρώτη ερώτηση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρήσαμε ότι θα προχωρούσε σε δημοπρασία. Περιμέναμε ότι θα ήταν γύρω στο 15 η τιμή ευρώ, ευρώ Άρα, πλέον δεν μιλάμε για 7 έως 8 δισεκατομμύρια, αλλά για 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο θέμα. Διαβάζοντας το έγγραφο επί του οποίου συμφωνήσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη με τη διαδικασία της επιτροπολογίας, στην ε, τη σκέψη υπαριθμών 11 αναφέρεται με σαφήνεια το εξή, προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνολογική ποικιλία τα προγράμματα ETS θα πρέπει να χρηματοδοτούνται. Και προγράμματα από 20 κατηγορίες ανανεώσιμων ενεργειών Σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη παριθμών 6, όπου αναφέρεται ότι 50% των project αυτών μπορούν να χρηματοδοτούνται, καταλήγει κανείς στον εξής αριθμό ένα πρόγραμμα CCS αντιστοιχεί σε 5 εκατομμύρια. Και αυτό θα σήμαινε 500 εκατομμύρια. 8 project θα σήμαιναν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά το θα μπορούσε να αφαιρεθεί για τη δέσμευση άνθρακα. Και αυτό φυσικά θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι μόνο 500 εκατομμύρια θα μένουν για νεονόσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή το 8πλάσιο, 10πλάσιο ποσό θα πήγαινε για τα συστήματα δέσμευσης άνθρακας από ότι για τα θέματα ε, για, για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ κατά δεύτερον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορείτε να μας ε, διαβεβαιώσετε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα υπάρξει τέτοια άδικη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των συστημάτων δέσμευσης άνθρακα, που παραπιπτόντως αποτελεί και ένα πολύ πιο δαπανηρό τρόπο και δεν είναι απόλυτα ουδέτερος ο τεχνολογικός, το τεχνολογικό αυτό μέσο ως προς ε, το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό ήταν πραγματικά μια άδικη κατανομή. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να κοιτάξουμε το άρθρο 8, παράγραφο 3 όπου αναφέρεται τα θέματα του συμψηφισμού. Θα πρέπει να σας το διαβάσω, συνάδελφοι, για να καταλάβετε τι εννοώ. Επειδή το συνολική... Αν οι συνολικές αντίσεις για χρηματοδότηση είναι πιο υψηλή από ότι τα κονδύλια, το οποίο είναι πιθανό, θα μειωθεί ο αριθμός των επιλεγμένων προγραμμάτων με την ίδια αναλογία για την κάθε ομάδα, με την ίδια δηλαδή αναλογία για τα συστήματα δέσμευσης άνθρακα και για τις ανανεώσιμες. Συνεχίζει λοιπόν το άρθρο και αναφέρει ότι όπου θα ε, επιλεχθούν τα φθηνότερα έργα σε ό,τι αφορά την τιμή δηλαδή ανατόνο. Άρα, έχουμε πολλά πιο πολλά κονδύλια ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συστήματα αποθήκευσης άνθρακα και πολύ, πιο πολλά προγράμματα, πολύ πιο πολλέ αιτήσει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς διασφαλίσετε λοιπόν ότι δεν θα πάνε όλα τα χρήματα στα συστήματα δέσμευση άνθρακα και δεν θα μείνουν τα ψηλά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοιτάξτε τους σχετικούς ε, ισολογισμούς. Γιατί τελικά δεν θα χρηματοδοτηθούν και οι πιο οι πιο άπορε ε, επιχειρήσεις, οι πιο μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ε, αν θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Τούρμες και στην περιγραφή του των ερωτήσεων ε, που τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγματι χρειάζεται να επιστρέψουμε εδώ στην οδηγία για το σύστημα εμπορία εκπομπών, όπου πράγματι ο νομοθέτης έχει προβλέψει Επιδοτήσει ε, ύψους 300 εκατομμυρίων, 300.000 ευρώ για, την, για αυτά τα δύο είδη έργων, δηλαδή έργων αποθήκευσης και δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα και έργων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, και πράγματι εμείς ανταποκρινόμαστε ε, πλήρως ε, στις διατάξεις και στο πνεύμα του νομοθέτη όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 10α εδάφιο 8. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Να τα απαντήσω επί τη ουσία Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δηλαδή το ζήτημα της ε, τιμή. Εμείς όπως γνωρίζετε δεν θέλουμε εδώ να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, ε, κοντολογίες, δηλαδή οι τιμές αυτές αντιδρούν με βάση την αγορά και πράγματι κάποιες εκτιμήσεις σήμερα μας λένε τα γύρω στα 300 εκατομμύρια βρίσκονται σε τιμή τώρα των 4 με 5 δισεκατομμυρίων πράγμα βέβαια το οποίο πάλι μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το ποιε είναι οι εκπομπές τώρα σε ό,τι αφορά την πώληση αυτών των περαιτέρω χρηματοδοτήσεων δηλαδή των 300 ε, εκατομμυρίων να σας θυμίσω ότι πρόκειται για διάθεσή του στη δευτερογενή αγορά Άρα λοιπόν μην τα συγχαίουμε εδώ με την ε, πρωτοβουλία, την ε, κύρια πρωτοβουλία αν θέλετε η οποία ήδη έχει περιγραφεί εδώ. Άρα λοιπόν αυτές οι επιδοτήσεις αυτές θα απολυθούν μέσα στην δευτερογενή αγορά νέα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία αναφέρεται και ρητά στην απόφαση και η οποία υιοθετήθηκε ως τέτοια με αυτήν δηλαδή την αναφορά από τα κράτη-μέλη. Η απόφαση λοιπόν προβλέπει ότι αυτές οι ενισχύσεις, αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν διατεθεί έως το τέλος του 2013. Και με αυτό το πνεύμα και με αυτό το σκεπτικό η απόφαση προβλέπει πως όλα αυτά τα έργα μέσα στην ε, προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να αποδείξουν ότι πράγματι θα μπορέσουν να έχουν ξεκινήσει να βρίσκονται σε λειτουργία έως τα τέλη του 2015. Άρα λοιπόν, ένα από τα κύρια ζητήματα ή μία από τις κύριες ανησυχίες οι οποίες ακούστηκαν. Να τις απαντήσω ως εξής η κατανομή, αν θέλετε, αυτών των ενισχύσεων σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα αφενό και τη ανανεώσιμη πηγή ενέργεια αφετέρου, θα κριθεί με βάση τι ανάγκε επίδειξη. Γιατί εδώ μιλάμε για επίδειξη, demonstration των σχετικών τεχνολογιών και έχουμε προβεί σε ευρύ διαβουλεύσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλου του εμπλεκόμενου φορεί ε, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία και είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτές οι 34 διαφορετικές κατηγορίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 8 κατηγορίες των ε, ε, έργων ε, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα πράγματι θα ανταποκρίνονται στις σχετικές ανάγκες των κλάδων. Ε, πράγματι το κάθε έργο σε κάθε ένα από αυτούς τους κλάδους θα χρηματοδοτηθεί κατά 50% του σχετικού για το έργο κόστος. Και το σχετικό κόστος ορίζεται στις σχετικές κατευθυντήρες γραμμές και ορίζεται με τον ίδιο τρόπο για τους διαφορετικούς ε, τομείς, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο για τα έργα δέσμευσης διοξήτου του άνθρακα και με τον ίδιο τρόπο για τα έργα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν θα έχουμε εδώ αναλογία σχετικού κόστους και σχετική χρηματοδότηση δηλαδή του κόστους αυτού για τα 8 αφενός ε, προγράμματα CCS ασφαλούς ε, δέσμευσης και τα τέσσερα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ακριβώ θα είναι το κόστο, γιατί μιλάμε για έργα καινοτόμου χαρακτήρα, αλλά λοιπόν εκ των προτέρων δεν μπορεί κανένα να προβλέψει, να εκτιμήσει το κόστο και δεν νομίζω πω είναι απαραίτητο να το ορίσει κανεί εκ των προτέρων, ώστε να προβλέψει μια κατανομή των ε, σχετικών προβλεπόμενων ε, πόρων. Άρα λοιπόν, όποια και αν θα είναι η αναλογία, οι πόροι οι οποίοι θα διατεθούν στο μέλλον θα διατεθούν με αυτήν την αναλογία. Αυτή η αναλογία δηλαδή είναι αυτή που θα κρίνει τελικά το ποιο είναι το ακριβές ε, ποσό το οποίο θα διατεθεί αφενό ε, για την ε, δέσμευση και αφετέρου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ναι, η δική μου ερώτηση ήταν πολύ σαφή όμω. Εγώ ρώτησα πώ θα διασφαλίσετε την κατανομή μεταξύ δέσμευση διοξιδίου αφενό ανανεώσιμων πηγών αφετέρου απάντηση επιτροπής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί έχουμε 8 κατηγορίες τεχνολογίας και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες θα λάβουμε. Μπορεί να έχουμε δηλαδή περισσότερες προτάσεις για έργα από τον ε, χώρο των ε, ανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτή η ανισοκατανομία αν θέλετε μπορεί να αποβεί προ όφελο των ανεώσιμων πηγών ενέργεια. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε ποιε προτάσει θα υποβληθούν Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και γι' αυτό δεν είχαμε προτείνει ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των προτέρων συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ των δύο ερωτημένων. Δεν γνωρίζουμε ποιε προτάσει θα υποβληθούν και δεν γνωρίζουμε το κόστο των έργων που θα προταθούν. Δεν είμαι λοιπόν σήμερα στη θέση να σας ε, εκφράσω μια εκτίμηση ότι δηλαδή πράγματι θα έχουμε περισσότερε προτάσει ε, στον τομέα της ασφαλού δέσμευση ή περισσότερε προτάσει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ε, δεν έγινε σχετική πρόταση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχουμε και αντίστοιχε πληροφορίε στη διάθεσή μα. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει η πρώτη πρόταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την υποβολή προσφορών και τότε θα λάβουμε υπόψη μας όλε τι προτάσει οι οποίε θα υποβληθούν με βάση τα κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί, θα γίνει αξιολόγηση και έτσι θα αποφασιστεί τελικά το ποια έργα θα επιλεγούν. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ελπίζουμε πως θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και μόνο τότε θα είμαστε σε θέση. Ποιε είναι οι προτάσει, ποιες δηλαδή, ποια ε, χρηματοδότηση ζητείτε και ποια αναλογία θα εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έξι έχουν στήσει το λόγο. Ντέιβι, Γκροστέτ. Μισό λεπτό, περιμένετε. Μισό λεπτό, Κλόντου μέσα να οργανώσουμε τη συζήτηση. Ντέιβι, Γκροστέτ, Μαγκάβαν, Μπαζικούτ, Βεγκαρδίνη, Έστερ Ντελόγκ. Άλλος. Επιθυμεί κάποιο άλλο να λάβει το λόγο, κυρία Ντεμπρόιν. Εντάξει. Λοιπόν. Εννέα έχουν ζητήσει το λόγο. Δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν να απαντήσει και το τρίτο τμήμα της ερώτησής μου για να έχουμε όλες τις προφορίες και να είναι λίγο πιο σαφής από ό,τι υπήρξε μέχρι τώρα. Κύριε τύρμες, κοιτάξτε, οι συνάδελφοι πρέπει να λάβουν το λόγο και μετά διακόπτη πρόεδρος, μα λάβατε μία απάντηση. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, πάντως ε, είναι απάντηση. Τώρα η απάντηση απαιτεί και άλλη απάντηση. τα πράγματα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήμουν ο αρμόδιος ε, για το CCS δηλαδή, δέσμευση και ε, πριν από τρία χρόνια και ένα μήνα είχε πει το Συμβούλιο πως θα ήθελε 12 ε, έργα επίδειξης ε, έως το 2015 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα της ε, δέσμευσης δηλαδή. Και αναρωτιόμαστε πού είναι αυτά τα έργα επίδειξης. Εάν τελικά περάσει λοιπόν αυτό το έγγραφο τότε μιλάμε για τα τέλη του επόμενου χρόνου μέχρι τα οποία θα έχει αποφασιστεί η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν μετά η σχετική προθεσμία στο 2015 για εφαρμογή θα είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ε, πως ε, η χρήση των ορυκτελέων ε, γίνεται με αυξανόμενους ρυθμούς. Ακόμα και η Κίνα η οποία έχει ξεκινήσει διάφορα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Παρόλα αυτά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη χρήση Ε, σε ό,τι αφορά ε, το αέριο και πάλι χρειαζόμαστε τη ληστηρία και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά το ΣΥΣ πράγματι πρόκειται για μια προσέγγιση την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω. Και αυτή εδώ η Επιτροπή ήταν εκείνη η οποία είχε προωθήσει αυτή την ιδέα δηλαδή τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων επίδειξη μέσω αυτών των χρηματοδοτήσεων. Κάναμε τι σχετικέ προτάσει, απευθυνθήκαμε ε, στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο μα απάντησε μετά από κάποιου μήνε ναι, πρόκειται για μια καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα σα δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι χρηματοδοτήσει. 13 μήνε πέρασαν από τότε και τι έχουμε μπροστά μα έκτοτε κάποιο σχέδιο για το πώ θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Ο Κλοντ ε, ε έθιξε κάποια πολύ σωστά ζητήματα. Δηλαδή αυτά τα 300 εκατομμύρια θα, θα, θα αξιοποιηθούν με τον ε, σωστό τρόπο για να μπορέσουμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε αντίστοιχα έργα και από τους δύο τομείς. Θα μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία του 2015 με βάση αυτήν την διπλή, αν θέλετε, προσέγγιση δηλαδή των δύο τομέων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα διασφαλιστεί αυτό. Και για να κλείσω με αυτό το σημείο, υπάρχει και μια ιδεολογική φύση συζήτηση, αν θέλετε. Ο Κλοντ είπε ότι όταν αυτή η πρόταση είχε έρθει στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2008 είχε λάβει την υποστήριξη όλων των ε, πλευρών. Αλλά όχι, δεν είχε την υποστήριξη των πρασίνων, ούτε καν είναι Λούκας. Ε, δεν, δεν συμφωνούσαν. Ε, δεν επιθυμούν πυρηνική ενέργεια, δεν επιθυμούν CCS. Δεν διόξιδη του άνθρακα. Άρα λοιπόν, Κλοντ, έθιξες κάποια έγκυρα εδώ ζητήματα, αλλά μην αγνοούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι ότι ιδεολογικά εσείς αντιτίθεστε σε αυτά τα έργα. Κυρία Γκροστέτ, αυτά τα οποία θα πω, Πρόεδρε, θα προσωμιάζουν με αυτά που είπε ο Σάρφος Ντέβις και εγώ υπήρξε συγγήτρια στην Επιτροπή Βιομηχανίας για την δέσμευση και ε, αποθήκευση του διοξείου του άνθρακα αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας. Ε, κοιτάξτε, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του πακέτου ενέργεια κλίματος για το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης. Ε, δεσμευθήκαμε σε ό,τι φορά τα πιλωτικά προγράμματα και χρηματοδότησή του. Θα πρέπει να πάμε μέχρι το τέλος. Ε, βρισκόμαστε στον τομέα της έρευνας. Ναι, είναι γεγονό ότι έχουμε ανάγκη αυτά τα ταμεία, πρέπει να πάμε μέχρι τέρμα. Ε, απόφαση ελήφθη. Δεν μπορούμε συνεχώ να αμφισβητούμε αποφάσει που λήφθησαν πριν από ένα ή δύο χρόνια. Δεν ε, είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν ε, ορισμένοι δεν είναι υπέρ των, ε, της χρήσης ε, άνθρακα, εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την Κίνα, αλλά ξέρουμε ότι και στην Ευρώπη χρησιμοποιούμε σε παραγωγή ρεύματο άνθρακα. και εκλείουν ε, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την χρήση του άνθρακα, δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσει και οι λύσεις αυτές ε, περνάνε μέσα αυτά τα επιλογικά προγράμματα. Χρειάζεται ω εκ τούτου να εξευρεθούν οι χρηματοδοτήσει ε, για να μην έχουμε μια ιδεολογική και ιδεολειπτική θέση. Ευχαριστώ κύριε Μαγκάμπανη. Παλιά με τον Κλόντ είχαμε συμφωνήσει σε πολλά ζητήματα, αλλά όχι σε αυτό. Και δεν ε, καταλαβαίνω για ποιο λόγο σε αυτό το στάδιο, ενώ είχαμε συμφωνήσει και ο Κρίς έχει δίκιο λέγοντας ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα CCS και να βρούμε κάποιο συμβασμό ε, και να προωθήσουμε τις ε, ανανεώσιμες πηγές. Αυτός ήταν ο συμβασμός που οποίο καταλήξει. Και τώρα η Κομισιόν που έχει εφαρμόσει αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, ε, εφαρμόζοντα την διαδικασία επιτροπολογία, θέλουμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο με πολιτικά επιχειρήματα. Εγώ είμαι υπέρ της δέσμευσης και της αποθήκευσης οι ε, επιχειρήσεις ε, χάλιβα εργάζονται για το πάνω στο ζήτημα αυτό της δέσμευσης και αποθήκευσης. Δίχως αυτή λοιπόν την ε, τεχνολογία δεν θα πρόκειται να πετύχουμε την ε, απαραίτητη μείωση ε, στην χρήση άνθρακα. Εάν αρχίσουμε λοιπόν να καθυστερούμε και να χρονοτριβούμε για μια ακόμα φορά, δεν πρόκειται να κάνουμε μια, να πάρουμε μια πόση προς την κατεύθυνση. Ναι. Ορισμένοι ανέφεραν ότι πολλές από τις ε, επιχειρήσεις ε, είναι ιδιαίτερα ε, ανθίζουσες, αλλά εντάξει αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα, εάν πρόκειται για μια πολιτική συζήτηση, την είχαμε την πολιτική συζήτηση, πήραμε την πολιτική απόφαση, η Κομισιόν εφάρμοσε αυτή την απόφαση και θεωρώ ότι η Κομισιόν σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει ποιο θα είναι το, ποιο είναι το κόστος του άνθρακα σε 10-15 χρόνια. Έχουμε και την οικονομική κρίση. Η Κομισιόν έχει δίκιο. 8 ε, κατηγορίες CCS και 30 κατηγορίες ανανεώσιμων. Εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την διαδικασία επιτροπολογίας αφού, αφού έχουμε ήδη νομοθετήσει, δεν νομίζω πως θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε στα θέματα Επιτέλου καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Γκαρντίν, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα επαναλάβω πράγματα που ήδη υπόθηκαν, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορούμε συνεχώς να ανοίγουμε κεφάλαια, να μπλοκάρουμε τα πράγματα και να μην προχωράμε, χωρίς να υπενθυμίσω ότι η απόφαση που λήφθη στο πλαίσιο της Επιτροπολογίας αντανακλά την επιθυμία τουλάχιστον 26 κρατών μελών και που στο τέλος έτυχε διαπραγμάτευσης για ένα χρόνο τουλάχιστον και πραγματικά αντανακλά ε, τις θέσεις ε, των κρατών και των κυβερνήσεων των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ακούμε τις <coughs> ενστάσεις των πράσινων συναδέλφων και θέλουν να επηρεάσουν μια εργασία που ήταν περίπλοκη, δύσκολη, αλλά και είναι κάτι το οποίο καθυστέρησε. Θα πρέπει να περάσουμε λοιπόν την νέες τεχνολογίες για να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ε, CCS για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε μια καθυστέρηση στην ε, επιστημονική απόδειξη ε, θα οδηγούσε σε περιβαλλοντικές καταστροφές. Τώρα, σε ό,τι φορά τι ενστάσει των συναδέλφων, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι υπάρχει η τελική σκέψη 11 τη υποζήτηση απόφαση, η οποία ρητά αναφέρει πως για να διασφαλίσουμε την ε, τεχνολογική ποικιλία θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε 8 προγράμματα πειραματικά CCS και ένα πρόγραμμα από τις υποκατηγορίες για τα ανανεώσιμες και στο παράδειγμα αναφέρονται 34 υποκατηγορίες ε, τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες ε, πηγές. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το σωστό, κάτι που απαντά στις ανησυχίες μας και θεωρώ ότι η τεχνολογία CGS είναι ένα πείραμα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε σύμφωνα με τα όσα αποφασίσαμε, διότι θεωρήσαμε ότι ανέκαθεν ε, την είχαν προτεραιότητα και είναι στρατηγική σημασία. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ του Άση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να διορθώσω αυτά που είπε ο Chris Davis για το παρελθόν, αν θέλετε, της πολιτικής αυτής απόφασης. Θα θυμάται ο Κρίς ότι ήμασταν αντίθετοι στην ιδέα να υπάρξει σύστημα υποστήριξης μόνο για το CCS. Ήμασταν όμως υπέρ της τελικής συμφωνίας που περιλάμβανε τα συστήματα αποθήκευσης άνθρακα συν τα συστήματα αποθήκευσης, ε, τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια όπως περιέγραψε πολύ σωστά ο Κλόντ. Και να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι σε ό,τι αφορά το πακέτο για το κλίμα που εγκριθήκε πριν από 2,5 έτη, υπήρξε η δυνατότητα να υποστηριχθεί de facto το CCS, ορίζοντας πρότυπα για τις εκπομπές κιλοβατώρα. τότε ο εισηγητής που ήταν υπεύθυνο για το CCS αποφάσισε να μην αγωνιστεί για την πολύ αυτή αποτελεσματική μορφή προώθηση του συστήματος CCS. Ευχαριστώ. Η κυρία Έστερ Ντελάνγκα, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση που έδωσε και νομίζω ότι εδώ είναι μια κλασική περίπτωση άρνησης των γεγονότων. Έχουμε τους μεν που υποστηρίζουν το σύστημα ETS ε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρει ότι συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα CCS αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να πω ότι όπως και οι συνάδελφοι μάλλον ε, έχω αμφιβολίες για την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να έχουμε διαφωνίες σε ό,τι αφορά τα ποσοστά. Μπορούμε να πούμε ότι το CCS, για παράδειγμα, είναι και πιο ακριβώς τεχνολογία, άρα είναι μάλλον λογικό να απορροφά πιο πολλά κονδύλια. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, θεωρώ, να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό σε ό,τι αφορά το ψήφισμα. Θεωρώ όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, θα πρέπει να κοιτάξουμε την πρόταση η οποία πήρε πάρα πολύ χρόνο μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας συνεχίσουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και σε επιταχύνουμε. Τελευταία παρατήρηση, ίσως και ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι στο διοξιδίου του άνθρακα είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο στόχος των δύο βαθμών. Γιατί πραγματικά αναρωτιέμαι πολλές φορές πόσο σοβαρά παίρνουμε το στόχο αυτό για τους δύο βαθμούς Κελσίου. Η κυρία um, Ευχαριστώ. Ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για το CCS τότε που διαπραγματευόμασταν το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια ο συνάδελφος που ήταν σκιώδης εισηγητής για το ETS, το σύστημα εμπορίας. Λοιπόν, και αυτός ε, υποστήριξε το ποσό αυτό των 300 εκατομμυρίων. Εγώ δυσκολευόμουν με το σύστημα CCS και ακόμα εξακολουθώ να δυσκολεύομαι σε ό,τι αφορά κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και θα έπρεπε να έχει καταστεί σαφές, θεωρώ, όπως είπε και η Σατουχάση. ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις τέτοιες για την Κίνα, για παράδειγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα χρήματα τα οποία δεν δαπανώνται για το CCS δεν πάνε απαραίτητα σε ανανεώσιμες πηγές μπορεί να πάνε σε παράδειγμα σε θέματα, σε τεχνολογίες άνθρακα ή πυρηνικής ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα τέτοια μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στη τελική ανάλυση χάρηκα που καταλήξαμε στη συμφωνία και όπως είπαν και οι πράσινοι, η συμφωνία προδιαγράφει με σαφήνεια και τη χρηματοδότηση του CCS και τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες. Αυτό ήταν το νομοθέτημα στο οποίο καταλήξαμε. Γι' αυτό λοιπόν να ρωτήσω το εξή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι δεν μπορούμε σήμερα να υπολογίσουμε την τιμή για το μέλλον. Συμφωνώ. Αλλά αν θέλετε να υπάρξει ισορροπία στο μέλλον, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει όντως αυτή η ισορροπία από τη στιγμή που τα έργα έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν σήμερα πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει αυτή η ισορροπία στη διαδικασία αυτή. Και μια δεύτερη ερώτηση. Στο τμήμα της οδηγίας που αφορά το CCS και όχι το ETS αναφέρθηκαν πολλές λεπτομέρειες για την περιβαλλοντική ασφάλεια. Μπορεί να μας διασφαλίσει, να με διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ότι αυτά τα πρότυπα, αυτά τα μέτρα ισχύουν και για τα έργα επίδειξη. Ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, χρειάζομαστε μεγαλύτερη ενεργεία από το τικότητα. Αυτό αποτελεί μια συνένεση εδώ και κατά συνέπεια χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Εκείνο το οποίο εγώ δεν αντιλαμβάνομαι είναι αυτή η συζήτηση να γίνεται αν θέλετε με ένα ιδεολογικά φορτισμένο τρόπο και να γίνεται ένα είδος αν θέλετε εδώ ταξικής επάλης ε, δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή αυτά τα ζητήματα εδώ δεν έχουν να κάνουν με το ερώτημα το οποίο καλούμαστε να επιλύσουμε το, το, πρόβλημά μας χρειαζόμαστε εδώ μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών λύσεων άρα ε, είτε το θέλουμε είτε όχι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτή την τεχνολογία του ΣΕΣ δηλαδή της δεσμευσικής αποθήκευσης δηλαδή με βάση και τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα και παντού, ε, νομίζω πως είναι σαφές ότι θα χρειάζεται να βρούμε μια τεχνολογία η οποία θα μας βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του διοξιδίου του άνθρακα, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα δηλαδή. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να έχουμε μια ε, σωστή ισορροπία αν θέλετε παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην υπάρχει καμία παραμέληση και εκείνου του τομέα. Εκείνο ε, ε, για το οποίο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν κινείται αντικειμενικά. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να μην να κάνει εκ των προτέρων εκτιμήσει και να προβεί σε μια δίκαιη κατανομή. Εγώ πιστεύω πω θα το πράξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με λυπεί πω ο, Κλοντ ε, Τούρμε, ένα ο οποίο είναι από του πλέον αποτελεσματικού εδώ, είναι τόσο κοντόθαλμο εδώ και πραγματικά θέλει με τόσο μονομερή τρόπο να αποκλείσει μία από αυτέ τι τεχνολογίε που μπορούν να μα βοηθήσουν εδώ. Εγώ ήθελα ή ήλπιζα ότι θα είχε παραμείνει μέσα σε αυτή τη γενική συνένεση που έχουμε επιτύχει. Δηλαδή και αυτό το σύστημα μπορεί να μας δώσει μια ε, μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούμε δηλαδή να, να, να, να εξασφαλίσουμε ε, ότι δεν θα υπάρχουν κάποιοι, ε, κάποια μέσα, δηλαδή κάποιες πηγές ενέργειας τις οποίες δεν θα λάβουμε καθόλου μα υπόψη, είτε αυτή είναι ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι πυρηνική ενέργεια, οτιδήποτε άλλο. ο Σπέτερ Λίζα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλά υπόθηκαν επί τη αρχή, γι' αυτό θα ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε εδώ να τσακωνόμαστε κατά πόσο χρειαζόμαστε ή όχι. Ε, εν πάση περιπτώσει έχουν υποθεί διάφορες ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο παγκοσμίω, αλλά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ε, χάλιβα, το τσιμέντο, είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να παράγουμε και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Χρειαζόμαστε δηλαδή εδώ ε, να και λύσει σε ό,τι αφορά και περαιτέρω ε, κλάδου οι οποίοι εμπλέκονται στον χώρο τη ενέργεια και θα ήθελα να ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο πράγματι λαμβάνει υπόψη τη και αυτού του τομεί τη δική τη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα εδώ κάποιου συναδέλφου ε, στην Επιτροπή που λένε ότι προβαίνουμε σε μια ιδεολογική ε, συζήτηση. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Δεν προβαίνουμε σε ιδεολογική συζήτηση. Και αν ακούσατε τον κλόν Τούρμε, δεν ξεκίνησε με δική του παρέμβηση μια ιδεολογική συζήτηση. Αυτό που ζήτησε ήταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία, ούτω ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση τόσο των έργων CSS, δέσμευση και αποθήκε, όσο και των έργων για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, ναι, δεν έχουμε στοιχεία ακόμα, αλλά έχουμε κάποιε εκτιμήσει. Και αν δούμε τι σχετικέ ε, τιμέ σε ό,τι αφορά το ε, διοξείδιο του άνθρακα, μιλάμε για 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει θέλει δίκαιη κατανομή μεταξύ CSS και ανανεώσιμων πηγών. Άρα λοιπόν τι ακριβώ σημαίνει αυτή η δίκαιη κατανομή. Στο επόμενο άρθρο μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξουμε καταρχήν 8 έργα CSS. Γνωρίζουμε επίσης πόσο ακριβά είναι αυτά τα έργα CSS. Άμα μιλάμε λοιπόν για 50% σύγχρηματοδότηση αυτών των 8 έργων CSS, μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρόκειται για ε, κάποιες εκτιμήσεις, οικοτολογίες από τον αέρα. Μιλάμε για συγκεκριμένες εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε με βάση τις τιμέ που ε, εκτιμούμε για το μέλλον. Άμα μιλάμε λοιπόν εδώ για 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δεσμευτούν από τις χρηματοδοτήσεις για τα έργα CSS και δεν περισσέψουν κονδύλια για όλα τα 34 λοιπόν υπόλοιπα έργα από τον χώρο των ανεώνυμων πηγών ενέργεια, ρωτούμε λοιπόν πώ θα διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή μεταξύ αυτών των κονδυλίων. Δεν είναι ιδεολογική συζήτηση. Σα παρακαλώ, στη συνέχεια κύριε Ντέβι, Σήμερα βρίσκομαι εδώ και ρωτώ ένα ερώτημα και αφήστε με, επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα. Ναι, θα θέλατε να είναι οδολογική συζήτηση, αλλά δεν είναι οδολογική συζήτηση. Είμαι ένα νέο ευρωβουλευτή εδώ, ρίχνω με ποιες αποφάσεις, δεν είμαι κατά του ΣΥΣΕΣ και απλά διακρίνω με βάση αυτά που έχω λάβει εδώ μπροστά μου ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ ένα μεγάλο κομμάτι, μια, ένα μεγάλο ποσοστό των κοντιλίων που έχουν δεσμευτεί για τη σηματοδότηση να πάει σε, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Άρα λοιπόν, εάν θέλει δίκαιη κατανομή μεταξύ αυτού του τομέα και των ανεμόσιμων πηγών ενέργειας, εγώ ρωτάω λοιπόν πώ θα διασφαλιστεί. Αυτό ρώτησε και ο Κλωτούρμε, αυτό ρωτάω και εγώ. Δεν λήφθη, σωστή απάντηση, σαφή απάντηση. Μα είπατε πω δεν θέλετε ε, να έχετε εκ των προτέρων δίκαιη κατανομή. Τότε μην το γράφετε. Μην γράφετε ότι θέλουμε δίκαιη κατανομή. Ή αλλιώ γράψτε το. Εάν δεν θέλετε πάντω, μην το γράφετε για να ξέρουμε, ναι, θέλετε εκ των προτέρων εσεί να διασμεύσετε, να δώσετε δηλαδή μέσω χρηματοδοτήσεων περισσότερα κονδύλια στο CSS. Εγώ, εκείνο εγώ που θέλω είναι να υπάρχουν απαραίτητα κονδύλια και για του δύο τομεί. Και για του CSS και για τι τι πηγέ ενέργεια. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν πρόκειται για λογική συζήτηση όπω θέλει να μα την παρουσιάσει ο κύριο Τέιβι. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν μήπω επιθυμεί να απαντήσει με σαφέστερο τρόπο στο ερώτημα που ετέθη. Εάν ναι, εντάχει, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να εξηγήσουμε κάπως περισσότερο πώς βλέπουμε το ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει παρανόηση σε ό,τι αφορά την φύση της απόφασης ε, που βρίσκεται στα χέρια των μελών του Κοινοβουλίου. Η τελευταία ερώτηση, από αυτή να ξεκινήσει σχετικά με την ισορροπία η απόφαση αναφέρει μια σειρά κατηγοριών ε, και για τα οποία μπορούν να υποβληθούν προγράμματα. Αναφέρθηκε ήδη πως έχουμε έκτο κατηγορίες για την ε, δέσμευση και την αποθήκευση και 34 για τις ανανεώσιμες ενέργειες. ενέργειας. Τώρα, τα αιτήματα για χρηματοδότηση, ας, ας υποθέσουμε ότι θα είναι 4 δις και για τα ανανεώσιμα πηγές, είναι 4 εκατομμύρια, τότε ε, θα δοθούν 50-50 οι χρηματοδοτήσεις. Όλα θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των προγραμμάτων που θα υποβληθούν, επιλέξιμα προγράμματα, προγράμματα που θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση. Είναι δύσκολο λοιπόν σήμερα να πούμε ποια προ... και πόσα προγράμματα θα υποβληθούν, πόσα προγράμματα θα αφορούν τα CCS και πώς ανανεώσουν πηγές ενέργειας, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα γίνει πρώτη επιλογή των CCS και μετά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, παράλληλα θα προχωρήσουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει καμία προτιμησιακή αντιμετώπιση. Σε Πάνω σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι ω Κομισιόν. Αυτό που λέμε εμεί είναι ότι έχουμε κάποιε απαιτήσει και για τι δύο κατηγορίε και για CCS και για τα ανανεώσιμα και σε αυτές τις δύο κατηγορίες ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ε, για προγράμματα τα οποία θα αξιολογηθούν. Περί αυτού η απόφαση είναι σαφέστατη και η απάντηση σχετικά με το ζήτημα της ε, ισορροπίας, εμείς δεν μιλάμε στην οδηγία για ισορροπίες, εμείς αναφέρουμε τι τεχνολογίες είναι και ποιες είναι επιλέξιμες Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη και που θα ζητήσουν χρηματοδοτήσεις για αυτούς τους μηχανισμούς. Τώρα, ποια θα είναι τα ποσά που θα δοθούν στη μία ή στην άλλη κατηγορία, αυτό είναι αδύνατο να υποθεί εκ των προτέρων. Το ζήτημα της ε, περιβαλλοντικής ακαιρεότητας ε, των προγραμμάτων CCS, ναι, θα διασφαλιστεί. Έχουμε μια οδηγία και η οδηγία εφαρμόζεται για όλα τα προγράμματα που περιέχονται στην απόφαση αυτή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβουμε αναφορά στην οδηγία. Η οδηγία εφαρμόζεται και όλα τα ζητήματα που άπτονται της προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη προστασία λαμβάνονται και αυτά υπόψη. Και τα προγράμματα CCS που θα επιλεγούν και θα υποστηριχθούν με βάση αυτόν τον κανονισμό δεν αφορούν μόνο θέματα παραγωγής ενέργειας. Ε, ασχολούμαστε και με άλλες όπως ε, το, τις ε, τις ε, και διάφορες άλλες βιομηχανίες. Η πρόεδρος ζητάει να ολοκληρώσει ο πρόεδρος της Κομισιόν να πω ότι όπως ορίζει το πακέτο για την κλιματική αλλαγή, όλα, ε, όλες οι τεχνολογίες ε, είναι χρήσιμες και οι δύο αυτές μας απασχολούν επίσης ε, πρόεδρος δεν χρειάζεται νομίζω να προβλέψουμε τροπολογίες θα ψηφίσουμε μεταξύ 26 και 28 Απριλίου και στην Ολομέλεια 17 με 20 Μαΐου Περνάμε τώρα στη διάσκεψη της Δόχα που δεν ήταν ε, και καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χεμπράντι για να μας ενημερώσει πλήρως αλλά και συντόμως. Και έπειτα θα περάσουμε στο ζήτημα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω τα αποτελέσματα τη Συνόδου τη Ντόχα ήταν μάλλον καταστροφικά. Από όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ε, λιγοστά μόνο πρέπει να πω ότι τελικά εγκρίθηκαν. Είδατε στην έκθεση, η οποία συντάχθηκε για την επίσκεψή μας ποια ήταν τα αποτελέσματα και πόσο άσχημα ήτανε. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν σήμερα το απόγευμα να εστιαστούμε σε κάποια πολιτικά ζητήματα. Καταρχά. είναι μάλλον ενοχλητικό το γεγονό ότι βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται τόσο πολύ στι ιστορικέ διαδικασίε για την εξέβρεση κοινή θέση και τελικά ξεχνάει ότι υπάρχουν 150 άλλα έθνη, χώρε στον κόσμο που είναι συμβαλόμενα μέρη του ΣΑΙΤΕΣ. Για παράδειγμα, λοιπόν, όταν καταλήξαμε στη συμφωνία για τον Ερυθρό Τόνο, ο Ιάπωνας υπουργό, ε, όσο καιρό εμείς κάναμε διαπραγματεύσεις, ε, πήγαινε σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, στην Αφρική, με ένα μεγάλο τσουβάλι χρήματα, για να εξασφαλίσει την ε, υποστήριξη της θέσης του για το παράδειγμα 1 σε ό,τι αφορά τον ερυθρό τόνο κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ντόχα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4-5 ε, ώρες κάθε μέρα διαβουλευόντουσαν για την κοινή τους θέση, μεταξύ τους δηλαδή. Αυτό φυσικά επηρεάζει την ε, επιρροή που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν σχεδόν μηδαμινή. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 ψήφους στην διάσκεψη ΣΥΤΕΣ, ενώ η Ιαπωνία, η Κίνα έχουν μόνο μία ψήφο. Άρα θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή αν επιλέγαμε μία διαφορετική προσέγγιση. Ένα άλλο πολιτικό ζήτημα είναι ότι το ΣΥΤΕΣ ε, στο παρελθόν αποτελούσε επιστημονική ε, συνάντηση όπου λαμβάνονταν επιστημονικές αποφάσεις. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Αποτελεί ένα πολιτικό φόρουμ και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν είναι κατάλληλα, αν θέλετε, για την λήψη αυτών των πολιτικών αποφάσεων. Το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας, το ΣΥΤΕΣ ήταν στο παρελθόν ένα από τα πιο αποτελεσματικά φόρα σε ό,τι αφορά τη ποικιλότητα και αποτελεί ένα από τα πιο, από τα λίγα που λαμβάνονται δεσμευτικέ αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο καταστροφικό το γεγονός ότι στην παρούσα φάση πολλά είδη τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και παράλληλα ακόμα και το ΣΥΤΕΣ δεν μπορεί να καταλήξει σε μία απόφαση. Και αυτό λόγω των βασικά των εμπορικών συμφερόντων. Κάθε φορά που υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα και αυτά παρεμβαίνουν, είναι δύσκολη η λήψη αποφάσεων. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις για κάποια φυτά, κάποια ε, δέντρα, αλλά όλα ήταν είδη τα οποία δεν αποτελούν είδη μεγάλης εμπορικής ε, σημασίας. Κάποιες χώρες όπως η Ιαπωνία ανέφεραν ότι πολλά ζητήματα για, τον, για κάποια είδη αλλιευμάτων δεν θα πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευση ε, στα πλαίσια της ΣΥΤΕΣ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα κοιτάξουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία αυτή για τον ερυθρό τόνο. Γιατί πλέον με τα καταστροφικά αυτά αποτελέσματα της Ντόχας θα πρέπει θεωρώ να επικεντρωθούμε στο θέμα της ICAD και να ασκήσουμε πιέσεις, ιδιαίτερα στους Κινέζους και στους Ιάπωνες, για να συμφωνήσουμε για τον ερυθρό τόνο στα πλαίσια της ICAT. Σας ευχαριστούμε. Ήσασταν σαφέστατος. Μπασικούτ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στα όσα είπε ο συνάδελφος, ο αγαπητός συνάδελφος Χαρμπράντη. Απλά να τονίσω τα δύο πολιτικά μηνύματα που μας εστάλησαν. Πρώτον, ότι καταρθώσαμε ως Ευρώπη να μιλάσουμε μία φωνή και μετά η Κοπενχάγη όλοι μας είπαν ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μιλούν με μία φωνή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα στην Τόχα, αλλά είναι ότι αργήσαμε να μιλήσουμε με μία φωνή. Δεν φτάσαμε καλά προετοιμασμένοι στην Τόχα και αγωνιζόμαστε να βρούμε κάποια κοινή θέση μεταξύ μας. Ε, η Κίνα και η Ιαπωνία είχαν ταξιδέψει και είχαν φροντίσει οι προτάσεις τους να γίνουν δεκτές στην Ντόχα. Εμείς μέσα σε δύο ώρες ιτηθήκαμε σε ό,τι φορά τον ερυθρό τόνο. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι θα πρέπει όχι μόνο να μιλάμε με μία φωνή, αλλά να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και η Κομισιόν να ε, λαμβάνει εντολή για τις διαπραγματεύσεις και να μην προσπαθούμε να βρισκόμαστε στις διασκέψεις αυτές 27 μέλη και να προσπαθούμε να συντονίσουμε την θέση μας την τελευταία στιγμή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθεί μετά από την συνάντηση της Δόχα διότι στην ε, Κανκούν θα υπάρξει διάσκεψη για το περιβάλλον τώρα. Το ζήτημα του ICAT, εδώ η Ευρώπη θα πρέπει να είναι συνεπής. Τελευταία συνάντηση της ICAT, εμείς δεν ήμασταν συνεπείς ό,τι φορά το αίτημα μας για τον Ευτροτόνο. Τώρα, ως Ευρωκοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να είμαστε κατά της ε, παράνομης εμπορίας ε, του ερυθρού τόνου, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτή η θέση θα ε, προωθηθεί και στο Παρίσι στην διάσκεψη της ICAT, διότι μέχρι τώρα η Ευρώπη έχει διαφορετική φωνή στην ICAT και διαφορετική στο CITES. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή μας θα είναι η αυτή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και την βιοπικιλότητα που αυτόν μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Μπαζίλ θέλει να λάβει το λόγο να μας πει κάποια πράγματα εντάχει. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι χρειαστήκαμε πολύ χρόνο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό μεταξύ μας, ενώ άλλα συμβαλόμενα μέρη στη διάσκεψη ε, επηρέαζαν τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να είμαστε στο μέλλον πιο αποτελεσματικοί τόσο στο πλαίσιο της ΣΥΤΕΣ όσο και στο πλαίσιο άλλων διαπραγματεύσεων στον χώρο του περιβάλλοντος. Δηλαδή το εν λόγω πρόβλημα αυτό δεν παρατηρείται μόνο στο πλαίσιο της διάσκεψης ΣΥΤΕΣ, αλλά σε πολλές ε, διαπραγματεύσεις έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις ε, για την ε, κύρωση της ε, τροποποίησης Γκαμπορών γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να αποτελέσει πλέον μέλος της διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια θα μπορεί να χρησιμοποιεί και τη δική της νομοθεσία για να ενδυναμώσει τη δική της θέση. Επίσης θα πρέπει να ε, συζητήσουμε το πώς θα μπορούμε να πείθουμε άλλα συμβαλλόμενα μέρη όταν συζητούμε ειδικότερα σημαντικά θέματα όπως για παράδειγμα ζητήματα αλληλεία ή εξηλεία. Πώς λοιπόν θα χρησιμοποιούμε σε σχέση με αυτά τα συμβαλόμενα μέρη με αυτέ τι χώρε, να χρησιμοποιούμε τα δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία, συμφωνή σύνδεση και καθεξή, ε, να χρησιμοποιήσουμε αν θέλετε το χάπι ε, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε ε, διατάξει στο πλαίσιο τη ε, Άρα λοιπόν αυτό το σκεφτόμαστε, αποκοινούμε το Κοινοβούλιο και σε σχέση με την ΑΚΑΤ και νομίζω πω ο Επίτροπο Ποτότσνικ θα θίξει αύριο εδώ το σχετικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε να λάβει το λόγο. Κυρία Κουτιέρες, πολύ σύντομα παρακαλώ. Είδα τα όσα συνέβησαν μετά από την Κομπεχάγη, θα πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Το ζήτημα δεν είναι να έχουμε μια ενιαία θέση στην Ευρώπη, αλλά είναι να είμαστε λογικοί και αυτό το οποίο προτείνουμε να είναι και εφαρμόσιμο. Εδώ όμως ε, προωθούμε έναν εθελοντισμό, ένα ιδανικό πνεύμα με εξαιρετικές προτάσεις, αλλά δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας. Θα πρέπει οι προτάσεις μας λοιπόν να είναι ρεαλιστικές και να γνωρίζουμε συνάμα το τι πιστεύουν οι άλλοι. διότι ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμες προτάσεις. Με ιδεολογίες δεν ε, κατακτάμε τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, στην προηγούμενη θητεία ήμουνα στην αντιπροσωπεία για, την ε, Ιαπωνική, το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο και ξέρουμε και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα δίγραφό της έκθεσης κάποια σχόλια προς την Ιαπωνική αντιπροσωπεία λέγοντας ότι όταν θα μεταβείτε στην, στο Τόκιο σας παρακαλούμε να θίξετε το θέμα αυτό και να ζητήσετε να το σκεφτούν. Ο κύριος Ναζέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση για τον ερυθρό τόνο απορρίφθηκε στην ΣΥΤΙΣ με 20 ψήφους ε, κατά 16 υπέρ. Αυτό τι σημαίνει ότι ο ερυθρός τόνος και πάλι επαφίεται στα πλαίσια της ICAD. Πρόκειται πραγματικά για μια καταστροφική, καταστροφικό αποτέλεσμα. Είχα θέσει στις 9 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο μια ερώτηση στην Ολομέλεια η οποία αντιμετώπιστε και ως ερετροϊκή ερώτηση. Γιατί είχα πει ότι δεν είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε μόνο κάποια ζητήματα, αλλά και για να καταστρώσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές. Δυστυχώς το αποτέλεσμα για τον ερυθρό τόνο μας δίταξαν ε, δύσκολα μαθήματα. Κυρία Γκροστέντ, Πρόεδρε, όταν διαπιστώνουμε τα όσα συνέβησαν στην Κοπενχάγη και στην Τόχα, μπορούμε να πούμε πράγματι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα αδύναμη και δεν κατορθώνει να ε, εισακουστεί σε διεθνέ επίπεδο. Εντάξει, εδώ στο Κοινοβούλιο μπορούμε να λαμβάνουμε ό,τι θέση θέλουμε, ό,τι μέτρα θέλουμε, αλλά δεν εισακόμεθα. Ε, απλούστατα διότι υπάρχουν 27 μέρη στο Συμβούλιο, 27 θέσεις ε, και όχι μία ενία και μοναδική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προκαταλάβουμε τα πράγματα, να μπορούμε να πείσουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, το δυνατόν αποτελεσματικότερες διεθνείς ε, διασκέψεις. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι με την άποψη αυτή. Και τώρα περνάμε σε ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό αφορά τα απόλυτα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φλόρεντς, για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είχα, το λέω ρεξί να πω κάτι σε σχέση με την Κοπεχάγη. Ίσως πραγματικά πρέπει να καλέσουμε εδώ κάποιους να μας πούνε ότι δεν α, α, λειτουργήσαν τα πράγματα στην Κοπεχάγη. Εν πάση περιπτώσει, ας περάσουμε εδώ στο τριπλή, όπως το λέμε. Είχαν ε, αποβληθεί εδώ κάποιες ε, τροπολογίες, είχαν γίνει κάποιες πολύ ε, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ήταν πολύ θετικό αυτό και με βάση τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί ε, βλέπαμε πως οι συνάδελφοι ε, συμφωνούσαν ε, με την προσέγγιση τη βασική που είχε ακολουθηθεί. Αυτές οι τροπολογίες ενίσχυσαν περαιτέρω τη δική μου θέση, άρα λοιπόν σίγουρα είναι συζητήσιμες μία σειρά από αυτές τις τροπολογίες και σε μία σειρά από προτάσεις θα μπορούσαμε πράγματι εδώ να δείξουμε μία διαλλακτική στάση εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχολιάσει ε, και τη σχετική στρατηγική. Για να είμαστε σίγουροι ότι τα όσα αξιώνουμε εδώ πράγματι θα μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Εγώ σας είπα ότι το δικό μου πεδίο εφαρμογής, εκείνο που επιθυμώ εγώ, είναι κάπως διαφορετικό γιατί ε, αρχικά είχαμε ονομάσει πολύ συγκεκριμένους τομείς και στη συνέχεια προβήκαμε σε κάποιες εξαιρέσεις. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν το πεδίο εφαρμογής θα έπρεπε να είναι πιο ευρύ αλλά δεν μπορούμε να το διευρύνουμε τόσο πολύ, ούτω ώστε ε, να έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο οικοδομικό μηχάνημα από τη μία πλευρά 50% τόνων, το οποίο να υπάρχεται σε σύντηση τάξη με έναν ε, ε, ηλεκτρικό, ηλεκτροκίνητο κινητήρα. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό πεδίο εφαρμογής θα πρέπει δηλαδή να ισχύσουν συγκεκριμένε εξαιρέσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ε, δημιουργούνταν νέα προβλήματα. Δεύτερο τώρα σημαντικό σημείο είναι το να κλείσουμε τις, ε, τα κενά εκείνα τα οποία καθιστούν δυνατές τις παράνομες εξαγωγές. Πρόκειται λοιπόν για ένα αποφασιστική σημασία σημείο. Ε, μιλάμε για μια εθνική αρμοδιότητα, άρα αντιλαμβανόμαστε πάλι πού εντοπίζεται το πρόβλημα εδώ σχετικά. Υπάρχει εδώ μια υποχρέωση ενημέρωσης, δηλαδή παροχής πληροφοριών που βαρύνει τους εξαγωγείς. Εδώ δηλαδή έχουν προβλεφθεί κάποιες αυστηρότερες διατάξεις, μπορούμε να τις ξανασυζητήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, εάν δεν μπορέσουμε να ελέγξουμε τις παράνομες εξαγωγές, τα ίδια τα σύνορα, Δηλαδή, εάν δεν δώσουμε τι κατάλληλε ιδεολογίε, τι οποίε δεν λαμβάνουμε μέχρι στιγμή οι τελωνιακοί μα υπάλληλοι τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντω, θεωρώ πω βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Μετά. Υπάρχει το ζήτημα τη αδειοδότηση σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το, πρόβλημα, το ζήτημα αυτό με προβλημάτισε αρκετά. Η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ένας ε, παραγωγός λαμπτήρων ο οποίος βρίσκεται δηλαδή άμεσα στα σύνορα με τις κάτω χώρες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε μια σχετική ε, δήλωση 27 φορές είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιθυμούμε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει καταχώρηση σε ένα κράτος μέλος και μετά ε, μέσω ενός συστήματος από κοινού ενημέρωσης πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών να επιτρέπουν την διάθεση σε όλα αυτά τα 27 κράτη-μέλη ε, του συγκεκριμένου λαμπτήρα ή της συγκεκριμένης τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται ε, για κάτι το οποίο ε, θίγει και την χρηματοδότηση, τις επιστροφές και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι τόσο απλό, αλλά να σας θυμίσω εδώ ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμά που εργάζονται ε, σε αυτή την Επιτροπή, σε αυτό το Κοινοβούλιο, επιθυμούν και τάσσονται υπέρ της ενιαίας αγοράς και ε, υπέρ της κατάργησης των σχετικών εμποδίων. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θέλουν να μην ισχύουν ε, οι ευρωπαϊκές διατάξεις σε ό,τι αφορά παλιές τηλεοράσεις και θέλουν να συνεχίσουν να ισχύουν εθνικές διατάξεις. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, βρίσκονται αν θέλετε λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ε, δηλαδή σκανδιναβικές χώρες και Αυστρία και μετά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη από τα αρχικα κρατημέλη μιλάμε δηλαδή από τα αρχικά 12 και από τα αρχικά 9 κρατημέλη που ε, έχουν πραγματικά πολύ άσχημες επιδόσεις σε αυτό το τομέα. Εν πάση περιπτώσει, όταν θα μπορέσουμε και όταν θα έχουμε καταφέρει να κλείσουμε τα σχετικά κενά και όταν οι εξαγωγείς θα μπορούν να τεκμηριώνουν πως ε, τα εν λόγω ε, προϊόντα εξακολουθούν να λειτουργούν, πραγματικά εξακολουθούν να λειτουργούν, τότε και το συνολικό ποσοστό του 65% είναι δυνατό. Αλλά αν υπάρχει ένα με δυο ένα ή δύο τέτοια παραθυράκια, αν θέλετε, στην νομοθεσία, τότε δεν θα μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Αν κλείσουμε τα κενά, δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε. Αυτό το Πώ βέβαια θα εκτιμηθεί το 65% ομολογώ πως είναι δύσκολο. Για παράδειγμα σε κάποιες χώρες όπως οι σκανδιναβικές ε, οι οποίες βρίσκονται εδώ και κάποιο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω μέλη και έχουν ε, ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης μπορούν πράγματι να παράσχουν αυτήν την τεκμηρίωση. Λέγοντας δηλαδή ότι ε, πρόκειται για το 65% των προϊόντων τα οποία διατίθεται στην αγορά. Αλλά για χώρες όπως η Βουλγαρία, και εδώ το εννοώ με καλοπρόεδρο τρόπο, δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Γιατί πολύ απλά και οι ε, σχετικές πωλήσει δεν, είναι, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να επιτρέψουν μια τέτοια εκτίμηση. Ε, στη Γερμανία, για παράδειγμα, σε τέτοιες χώρες μπορούν, ε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάποια κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ισχύσουν, για παράδειγμα, πόσα τέτοια ηλεκτρικά προϊόντα περιλαμβάνονται στα απόβλητα. Είναι ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, αλλά ποιο τελικά θα το ορίσει, ποιο μπορεί δηλαδή να υπολογίσει αριθμητικά ε, πόσα, ε, πόσες τέτοιες ηλεκτρικέ συσκευές θα στα απόβλητα. Για παράδειγμα στην Αυστρία ε, μου είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό να γίνει με σοβαρό τρόπο, με αξιόπιστο τρόπο. Γιατί βέβαια οι επιχειρήσει εδώ ε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά δηλαδή τα ποσά τα οποία θίγονται εδώ. Άρα θα πρέπει να είναι σοβαρές αυτές οι εκτιμήσεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας προτείνει ένα τρόπο, μια μέθοδο η οποία θα οδηγήσει σε μια καλύτερη θέση και τα νέα κρατημέλη, ναι, θα συμφωνούσα. Αλλά θα πρέπει να μου το εξηγήσει, να λάβω και κάποιες εξηγήσεις στο πώς θα λειτουργήσει αυτό. Άρα λοιπόν οι ε, τροπολογίε του συναδέλφου Σέβασε, εντάξει δεν λέω ότι διαφωνώ με αυτέ, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πώ θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Έχουμε για παράδειγμα ένα ε, παιχνίδι ε, στην ευρωπαϊκή αγορά, γνωρίζουμε το τι ισχύει, ποια είναι η τιμή και ό,τι καθεξής. Αυτά μπορούν να γίνουν σωστά. Αλλά σε ό,τι αφορά τους λαπτήρε, οι οποίοι για παράδειγμα χρησιμοποιούνται σε μια αποθήκη ή ε, φυλάσσονται κάπου, ε, πώς μπορούν να γίνουν σχετικές εκτιμήσεις δεν ξέρω. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας απαντήσει. Πόσο ρεαλιστική δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια τέτοια εκτίμηση. Εάν μπορούμε να γνωρίζουμε, ναι, τόσες συλλεκτικές σεβές στα απόβλητα, ναι, τότε μπορεί να είναι ένα τέτοιο σύστημα πιο αξιόπιστο, πιο ε, σοβαρό και πιο εύκολο στην εφαρμογή, πιο απλό. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, εδώ κατ' εξαίρεση είμαι λίγο πιο συντηρητικός, ε, θεωρώ δηλαδή πως και η κοινωνία και ο πολίτης έχει να αναλάβει εδώ μια ευθύνη σε ό,τι αφορά τις, ε, ε, τις παλιές τις Ε, το να έχουμε δηλαδή σημείο συλλογή ε, στην ίδια την επιχείρηση, το οποίο βρίσκεται και εγώ δεν ξέρω πού, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξεπεράσουμε λίγο. Δηλαδή χρειάζεται και ανάληψη ευθύνη από την κοινωνία και τον πολίτη. Όχι απευθείας καταβολή αν θέλετε του τέλους από τον πολίτη αλλά για μας για πώς το κάνουμε η ίδια η κοινότητα, ο Δήμος δηλαδή συλλέγει τις παλιές συσκευές μία φορά το μήνα και μέσω λοιπόν εγώ ως πολίτης μέσω του Δήμου της κοινότητάς μου καταβάλω το σχετικό αν θέλετε τέλος για την συλλογή αυτών των ε, παλαιών ε, συσκευών ε, και εντάξει πραγματικά τίποτα <laughs> δεν είναι δωρεάν ε, σε αυτή τη ζωή. Ο καθένα δηλαδή θα πρέπει να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, το αντιλαμβάνομαι. Ε, κάποιοι τώρα συνάδελφοι επιθυμούν να υπάρχει ένα ποσοστό ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση δηλαδή, ε, σε ό,τι αφορά τι συσκευέ. Ε, εδώ νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε μια συγχώνευση αν θέλετε των σχετικών ποσοστών, δηλαδή ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησης. Εγώ συμφωνώ με μια τέτοια προσέγγιση, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι επιθυμούν ε, ξεχωριστά αυτά τα δύο τα ποσοστά. Γύρω στο 5% νομίζω είναι η αξίωση των συναδέλφων. Ε, εγώ μπορώ να δεχτώ και αυτή την προσέγγιση, αλλά εάν αποφασίσουμε να έχουμε ξεχωριστά ποσοστά, τότε για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να πούμε, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, ότι ε, οι φορεί εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να προβούν σε μια τέτοια επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να έχουν μια, στη διάθεσή τους αυτές τις συσκευές. Δηλαδή Εάν ε, μαζέψει κανείς όλες αυτές τις συσκευέ ε, και μετά υποστούν αυτές μια μεταφορά η οποία τις καταστρέψει όλες και δεν μείνει τίποτα, τότε πραγματικά πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα πρέπει να ε, προβλεφθεί και κάτι αντίστοιχο αν θέλουμε ξεχωριστό ποσοστό για την επαναχρησιμοποίηση. ευχαριστώ. Θα σταματήσω εδώ για να μην περιλαμβάνω και περισσότερες εργασίες για τον εξαιρετικό μα πρόεδρο. Ε, άρα λοιπόν μπορώ να συμφωνήσω με την πλειοψηφία των ε, τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Κάρα Φλόρεντς ε, για την αποτελεσματική του εδώ συμπερίληψη διαφόρων τροπολογιών. Έχουμε 5 με 10 5 με 10 λεπτά καθυστέρηση. Άρα λοιπόν οι σκιώδεις συζητητέ θα πρέπει να λάβουν το λόγο για μόνο 3 λεπτά και οι υπόλοιποι ομιλητές μόνο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό όριο. Η κυρία Φαμπρέμπτο, όπως είπε ο, ο εισηγητής, ε, υποβλέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες σε μια πολύ καλή έκθεση και το τονίζω αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η εισηγητής έκανε κάποιες κινήσεις που ενισχύουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οποίες στηρίζουμε εμείς από την ομάδα μας. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστούν περαιτέρω. Το πρώτο, και το ανέφερε και ο εισηγητής, χαίρομαι που ε, είπε ότι επιδεικνύει ανοιχτό πνεύμα, είναι το θέμα της επαναχρησιμοποίησης, ε, το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε με τη θέση ξεχωριστού του στόχου, αλλά και διασφαλίζοντας ότι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην επαναχρησιμοποίηση αυτή θα πρέπει να ε, έχουν γρήγορη πρόσβαση στον κύκλο αυτό. Αυτό που ανέφερε και ο εισηγητής. Και τρίτον, να διασφαλίσουμε ότι θα διατίθενται γρήγορα πληροφορίες σε αυτούς που θα πρέπει να μεταχειρίζονται τα προϊόντα αυτά. Μία δεύτερη σημαντική γραμμή την οποία θα συζητήσουμε μεταξύ των ομάδων αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως είναι ποιοι είναι οι στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να προβληθούν και πώς θα πρέπει να υπολογιστούν αυτή η συζήτηση που αναφέρεται για τα οικονομικά προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί στην αγορά ή για το πραγματικό ύψος των ε, αποβλήτων στην αγορά. Εμείς από πλευρά της ομάδα μας υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες και συμφωνήσαμε με την συνένεση που φαίνεται να επικρατεί μεταξύ κάποιων ε, παραγωγών όπως ε, η Digital Europe και του Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Περιβάλλον σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες ροές αποβλήτων. Αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν και πολλά καλά επιχειρήματα για άλλες ε, προσεγγίσεις. Άρα και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κατά τρίτον, η προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στις μικρές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά ε, αποτελούν και σημαντικό τμήμα των συνολικών αποβλήτων, για παράδειγμα ε, παιχνίδια, ηλεκτρικές οδοντόβουτσες, ε, κινητά. Πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνουν πολύτιμα υλικά. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε αυτά και να τα υπογραμμίσουμε στην οδηγία προκειμένου και αυτοί, αυτές οι μικρές συσκευές να συνοδευτούν από ειδικού στόχους και να επικεντρωθούμε στην συλλογή και την ανακύκλωση αυτών των μικρών αλλά πολύτιμων συσκευών. Η συζήτηση μετά για τον σχεδιασμό των προϊόντων και την μεμονωμένη ευθύνη των παραγωγών. Νομίζω ότι εδώ πέρα επικρατεί γενικά ε, συνένεση στην Επιτροπή μας. Αν παράγει κανείς δύο υπολογιστές και ο ένας παράγεται με το χ τρόπο προκειμένου να είναι εύκολα ανακυκλώσιμος, αυτό δεν είναι σωστό μόνο από πλευράς marketing, αλλά θα πρέπει να συνεπάγεται και χαμηλότερη τιμή για την απόρριψη του προϊόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε στην οδηγία αυτή. Και αυτές είναι οι γραμμές που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Αν μου επιτρέπετε να θίξω και ένα τελευταίο σημείο, εν συντομία Πρόεδρε. Πολλές τροπολογίες υποβλήθηκαν, όχι από την ομάδα μας, αλλά και από άλλες ομάδες, για να μην συμπεριληφθούν τα ηλιακά πάνελ στην οδηγία. Αυτό πραγματικά με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί είμαι υπέρ των ε, ηλιακών πάνελ και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν έτσι εύκολα από την οδηγία. Και θεωρώ ότι τα σχετικά, οι σχετικές διατάξεις δεν ε, είναι αντίθετες και πολύ, πολύ λυπάμαι που δεν έχω περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Κρις Ντέιβις για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι γενικά σωστά εφαρμόζει και καλά εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, δεν τα πάμε και άσχημα, αλλά δεν είμαστε και τόσο καλοί όσο νομίζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ναι, ναι, θα φτάσω και σε αυτό που λέτε. Σχόλια εκτό μικροφώνου. Κάποιε φορέ η νομοθεσία από τι Βρυξέλλε φτάνει στο Λονδίνο και στο Λονδίνο την εξετάζουμε και μα φαίνεται ότι είναι από το διάστημα. Και αντί να κοιτάξουμε στην Ευρώπη να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται ε, αυτές οι νομοθεσίες κάπου αλλού στην Ευρώπη και κατά πόσο υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, αποφασίζουμε να επανεφεύρουμε πάντα κάθε φορά τον τροχό. Και φυσικά το αποτέλεσμα είναι πάντα απογοητευτικό. Και αυτό ισχύει και με την νομοθεσία αυτή. Γιατί στην αρχή όλοι υποστηρίξαμε την αρχή της ευθύνης του παραγωγού και η ενιαία αγορά όπως είπε ο Καλ Χάιντς, αποδεχόμαστε και προσυπογράφουμε την ιδέα ότι η παραγωγή τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσουν ότι η παραγωγή, οι τρίτοι φορείς που ενεργούν εκ μέρους τους θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας για τη σωστή ανακύκλωση των προϊόντων. Μπορεί να θεωρούμε ότι είναι αρκετά σαφής αυτή η διατύπωση, η παραγωγή, τα τρίτα μέρη. Αλλά τι λείπει εδώ είναι ο σύνδεσμος, η σύνδεση με τους παραγωγούς. Άρα επιτρέπουμε ουσιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους να συλλέγουν τα προϊόντα, να τα παρατάνε στους παραγωγούς, οι οποίοι μετά καλούνται να πληρώσουν το κόστο αυτό. Είτε πιστεύουν ότι το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό συλλογή είναι αποτελεσματικό ή όχι. Άρα θα ήθελα έναν απλό ορισμό, ο οποίος θα ξεκαθαρίζει ότι τα τρίτα μέρη τα οποία δρούν εξ ονόματος των παραγωγών θα πρέπει και αυτά να ορίζονται από τους παραγωγούς. Θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση για να υπάρχει σωστή απόδοση ευθυνών α, των, στους παραγωγούς και όχι εκμετάλλευση των παραγωγών αυτών. Και τέλος, ελπίζω να διασφαλίσουμε ότι όταν περάσει αυτή η νομοθεσία θα έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της εξαγωγής των αποβλήτων σε άλλες χώρες όπου δεν θα πρέπει να εξάγεται. Ο Καλ Χάιντς ε, θα πρέπει, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική τέτοια προϋπόθεση. Έχω υποβάλει μια τροπολογία σχετικά και ζητώ να υπάρξει πιστοποίηση, να υπάρχει επισήμανση για κάθε προϊόν. Θα πρέπει κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη τη λειτουργή το κάθε προϊόν. Είναι σωστή η αρχή που υποστηρίζει ο Καρλ Χάιντς. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση. Θα πρέπει το κάθε προϊόν το οποίο προορίζεται για εξαγωγή να διασφαλίζεται ότι λειτουργεί. Ευχαριστώ κύριε Στραμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς, ε, όπως είπαμε και την άλλη φορά, Είδαμε την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ε, εξοπλισμού ως μια σημαντική ευκαιρία για πιο αποτελεσματική τόνωση του οικολογικού σχεδιασμού των σχετικών προϊόντων, για τόνωση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και για ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στην τιμή των προϊόντων, ζητήματα στα οποία δεν ήταν ικανοποιητική η φυστάμενη οδηγία. Καταθέσαμε λοιπόν μια σειρά τροπολογιών για να μην περάσει να η ευκαιρία αυτή. Η πρόταση οδηγίες Επιτροπής βελτιώνεται ακόμη περισσότερο αν δώσουμε έμφαση στους παρακάτω τομείς. Την έμφαση της, της εξασφάλισης της εφαρμογής της αρχής της υπευθυνότητα των παραγωγών, ώστε αυτοί να καλύπτουν το πλήρες κόστος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ακόμη, την ε, υιοθέτηση πιο συγκεκριμένων και φιλόδοξων στόχων συλλογής, την υιοθέτηση ενός στόχου 5% λέμε εμείς για την επαναχρησιμοποίηση, την αποφυγή διαρών εξοπλισμού από την επίσημη και την προβλεπόμενη αλυσίδα και την παραπέρα διερεύνηση για περιεκτικότητα σε νανοηλικά, nanomaterials των ε, αποβλήτων αυτών. Αν και η έκθεση Florence ε, κάνει βήματα ε, προς αυτές τις ε, κατευθύνσεις, μένουν αρκετά τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπληρωθούν με τις τροπολογίες. Η έμφαση στην ευθύνη του καταναλωτή υποβαθμίζει το ρόλο των διανομέων και αγνοεί την ανάγκη για πόρους που έχει η αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε επομένω πως οι διανομείς θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο και πέρα από την πρακτική της ανταλλαγής παλιάς και νέας συσκευής για παράδειγμα μέσα από την απέτηση ειδικού αποθηκευτικού χώρου ε, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού για διανομής ενός μεγέθους και άνω και την υποχρέωσή τους να λειτουργούν και ως σημείο συλλογής τουλάχιστον για μικρές συλλογές, ε, συσκευές. Ταυτόχρονα να απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πόρους προς την αυτοδιοίκηση για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και βελτιστής ε, λειτουργίας των συστημάτων συλλογής θεωρούμε σημαντικό να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η αποκομιδή εξοπλισμού από τον οικοκυριά. Σχετικά με τους στόχους συλλογή, η οδηγία πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική με πρόβλεψη για συγκεκριμένους στόχους, για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που είναι πιο πιθανό να οδηγούν σε ταφή όπως οι λαμπτήρες και οι μικρές συσκευές. Επίσης είναι σημαντικό να απαιτούνται πληροφορίες για τα παραγόμενα των μονάδων ανακύκλωσης και όχι μόνο για τις ποσότητες που στέλνονται για ανακύκλωση προκειμένου να μετράται η πραγματική συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση καταθέτουμε τροπολογίε που αναφέρονται συγκεκριμένα στην προτεραιότητα τη επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης σε σύγκριση με την καύση. Ε, και σχετικά με την παρακολούθηση των ροών του εξοπλισμού και προκειμένου να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα κάθε τμήματος της αλυσίδας προτείνουμε τη συλλογή πληροφοριών εισόδου-εξόδου σε κάθε τέτοιο τμήμα. Ομοίως πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση των φορτίων εξοπλισμού προς επιδιόρθωση και παραγωγή αντίστοιχων αναφορών. Το Ευρωκοινοβούλιο Πιστεύουμε πως πρέπει να ζητά από όλα τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά σχέδια βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων αυτών με αναφορά και αξιολόγησή τους. Και τέλος επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε με νομικά δεσμευτικό τρόπο τις εξαγωγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε στις διάφορες εδώ τροπολογίες ε, υπάρχει εδώ μια σύγχυση, δηλαδή μια πληθώρα διαφορετικών ιδεών ε, σε ό,τι αφορά τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε, σε ό,τι αφορά τη συλλογή ε, Και εκείνο που θα ήθελα εγώ να επιτύχω και με την τροπολογία μου αυτό προσπαθώ να κάνω, είναι να να έχουμε διαφορετικούς στόχους συλλογής για διαφορετικά είδη, αν θέλετε, ε, δηλαδή έχουμε διαφορετικά, διαφορετικούς αριθμούς που μας προκαλούν σύγχυση για ε, διαφορετικά προϊόντα. Για παράδειγμα πετάμε το πιστολάκι για τα μαλλιά συνήθως στα απόβλετα, στα σκουπίδια, αλλά συνήθως ανακυκλώνουμε δηλαδή δίνουμε πίσω και παίρνουμε καινούριο κινητό τηλέφωνο και θα πρέπει να διευκρινίζεται ε, εδώ το γιατί συμβαίνει αυτό και θα θέλαμε να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι δική της άποψη. Συμφωνεί δηλαδή με το να θεσπιστούν διαφορετικά ποσοστά για διαφορετικά είδη προϊόντων. Επίσης, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμπεριφοράς του καταναλωτή, θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τη σημασία του να εξεταστούν τροπολογίες οι οποίες καλούν ή αξιώνουν καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή γιατί ε, νομίζω πως δεν αντιλαμβάνονται ακόμα πλήρως τι ευθύνε ε, που του βαρύνουν και δεν διευκρινίζεται αυτό με τον σωστό τρόπο σε διάφορα κράτη-μέρη. Αλλά λοιπόν θα πρέπει να ε, το ρυθμίσουμε και αυτό και επίση θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παράσχουμε κίνητρα στους καταναλωτές να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Είναι όλα ωραία το να κάνουμε λόγο για την ευθύνη του καταναλωτή, αλλά εάν δεν το πράττει τελικά ο καταναλωτής, δεν είναι επειδή είναι κακός άνθρωπος, αλλά είναι επειδή δεν αντιλαμβάνεται πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς ε, μπορεί να κάνει μια διαφορά από τη δική του πλευρά και ό,τι καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παράσουμε στον καταναλωτή τόσο τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο και ένα χάρτη πορεία αν θέλετε, ένα roadmap για το τι θα κάνει για να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Όχι απλά κάποιε γενικέ ιδέε. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από τροπολογίε, οι οποίε θα μα επέτρεπαν να επιτύχουμε ακριβώ αυτό και θα κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντα ότι εδώ δεν θέλουμε μόνο να έχουμε συγκεκριμένου στόχου, αλλά θέλουμε να έχουμε και έξυπνου στόχου, δηλαδή ευέλικτου στόχου και στόχου οι οποίοι θα είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζαμπίνεβιλτ. Εμείς υποβάλαμε 10 ε, τροπολογίες με στόχο την ε, συλλογή όσο γίνεται περισσότερων παλαιών συσκευών ώστε να μην ε, υπάρξει εξαγωγή τους ε, με αποτέλεσμα δηλαδή να έχουν πλαβερές συνέπειες σε ανθρώπους και το να καταλήξουν κάπου σε κάποιες χωματερές. Να πούμε τώρα κάτι, συγκεκριμένα, κάτι συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά το 65% των νέων πολλούμενων συστημών και του σχετικού στόχο, θεωρούμε πως ε, δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικός, γιατί η ε, παραγωγή, εκείνο το οποίο θα πράττουν, είναι, ε, θα είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των βαρέων συσκευών όπως πλυντήρια, για να επιτύχουν αυτό το ποσοστό του 65%, ενώ όλε άλλε άλλες μικρότερες συσκευές όπως είναι τα τηλέφωνα και ούτω καθεξή, δεν θα συλλέγονται, παρότι αυτά ακριβώς τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν περισσότερες ευλαβαρές ουσίες. Άρα λοιπόν καθώς ο κλάδος δεν έχει ανταποκριθεί και με τον κατάλληλο τρόπο έχουμε υποβάλει τις αντίστοιχες τροπολογίες. Άρα λοιπόν εμείς ε, θέλουμε να έχουμε 85% ποσοστό και ο συγκεκριμένος υπολογισμός να γίνεται ανακατηγορία προϊόντος. Επίσης ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία σε ό,τι αφορά τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών ε, τις τεχνολογίες δηλαδή IT να έχουμε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων γιατί τα εν λόγω εδώ προϊόντα διατρέχουν μια πολύ, ε, με πολύ μεγάλη ταχύτητα τεχνολογικές καινοτομίες με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος ρυθμός αντικατάστασής τους και κατά συνέπεια ε, θα μπορούσε να, υπάρχει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για τους ε, κατασκευαστές ώστε να είναι ε, πιο ανακυκλώσιμα, πιο εύκολα ανακυκλώσιμα τα προϊόντα τους και υπάρχουν μια σειρά από μεγάλους ομίλους οι οποίοι κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θέλουμε να υπάρχει και ευθύνη ε, των κατασκευαστών με βάση δηλαδή την αρχή εκείνου το οποίο το προκαλεί, δηλαδή για την φύλαξή τους, για την επαναχρησιμοποίηση και ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, είναι, ε, να προβλέψουν το, και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει, υπάρχουν κατάλληλα σημεία διανομής και κατάλληλοι μηχανισμοί ε, συλλογής και επίσης έχουμε υποβάλει μια περαιτέρω τροπολογία η οποία εστιάζει στην μηχανική επεξεργασία των παλαιών συσκευών. Ήδη δηλαδή από το πρώτο βήμα αν θέλετε της ε, διαδικασία επεξεργασίας θα πρέπει να απομακρύνονται οι βλαβερές ουσίες από αυτά τα προϊόντα και στη συνέχεια θα πρέπει να περνάνε από ε, περαιτέρω επεξεργασία τα προϊόντα. Ε, άρα λοιπόν η κοπή αν θέλετε σε πολύ μικρά κομμάτια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευθεί. Συνήθως δηλαδή με βάση αυτή τη διαδικασία της κοπής δεν γίνεται ακριβώ αυτό ο διαχωρισμό των πλαβερών ουσιών, πράγμα το οποίο δεν επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να περάσουμε στου υπόλοιπου ομιλητέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Καλ Χάιντ, ο κ. Σέπερ, για την ε, εξαιρετική έκθεση και για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδεξε, το οποίο ξεπερνάει τα όρια της, ε, των ομάδων. Σχεδόν σε όλα σύμφωνο μαζί του. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία με βρίσκουν, ε, έχω διαφορετική ε, θεώρηση η Αυστρία σε πολλές περιπτώσεις ότι έχει διαφορετικά συστήματα συλλογής και άρα με την πρόταση αυτή θα τεθούν σε εφαρμογή διατάξεις οι οποίες στη θεωρία μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ καλές αλλά από πρακτικής άποψης και από πλευράς νομικής εφαρμοσιμότητας δεν μπορούν ακόμη να εφαρμοστούν. Γιατί κοιτώντας τον ορισμό του Ευρωπαίου παραγωγού και της ευθύνης τους που προτείνει ο Καλ Χάιντς, ε, πολύ απλά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κοινότητα και το κόστος θα πρέπει να αναλυφθεί από τον παραγωγό ή αυτόν που διαθέτει για πρώτη φορά το προϊόν στην αγορά. Όσο έχουμε λοιπόν διαφορετικά συστήματα τα οποία ισχύουν, θα πρέπει να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις. Νομίζω όμως ότι βρισκόμαστε στο σωστό ε, δρόμο σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις συλλογής. Ε, καταλαβαίνω ότι και δέχομαι το 65% αλλά ως ποσοστό βάσης. Δεν νομίζω ότι θα ήταν το σωστό κριτήριο. Ίσως θα έπρεπε στα πλαίσια της επιτροπολογίας να εξευρεθεί ένα διαφορετικό σύστημα. Για παράδειγμα, να δούμε τι ποσοστό ηλεκτρικών αποβλήτων περιλαμβάνεται στα απόβλητα. Θα πρέπει να το εξετάσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ σε ό,τι αφορά την παράνομη αποστολή θα πρέπει να ισχύουν αυστηρές ρυθμίσεις και να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον τίθενται αυστηρές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριος Κυλακάκης. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό. Έχουν ε, γίνει πολύ καλές τροπολογίες και η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο δύο μικρές τροπολογίες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι χρήσιμες. Η πρώτη αφορά τους λιανεμπόρους, οι οποίοι θα πρέπει να συνδράμουν και σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση αλλά και σε ό,τι αφορά τη συλλογή μικρών συσκευών με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν θα εμπλέξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο τους μεγάλους ε, λιανέμπορους και θα βοηθήσει γιατί θα δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά πολλές συσκευές. Δεύτερη τροπολογία που προτείνω αφορά τα κράτη-μέλη και τη δυνατότητα που έχουν για επιπρόσθετα συστήματα για έναν σωστό τρόπο, για ένα κουπόνι αντιμετώπισης με οικονομικό τρόπο των ε, αποβλήτων αυτών. Τα κουπόνια αυτά θα ισχύουν σε περίπτωση όπου η παραγωγή χάνουν μεγάλο τμήμα των αποβλήτων και πρόκειται για πολύτιμα απόβλητα τα οποία δεν φτάνουν στα χέρια των παραγωγών. Βγαίνουν εκτό ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο οικονομικό κίνητρο και αυτό το κουπόνι αποτελεί ένα τέτοιο οικονομικό κίνητρο και αποτελεί και περαιτέρω ένα κίνητρο για την ανακύκλωση. Η τροπολογία επαριθμών 201, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές ήταν οι δύο τροπολογίες που είχα να προτείνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, κυρία Μερκής. Ε, ναι, είναι καλή ρύθμιση αυτή μετά την έγκριση κάποιων τροπολογιών θα βελτιωθεί περαιτέρω. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σωστοί στόχοι, αλλά και κυρίως ρεαλιστικοί στόχοι. Και συμφωνώ ιδιαίτερα με την κυρία Κατλέν Φανμπρέντ ότι και τα ηλιακά πάνελ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν από, την, από το νομοθέτημα αυτό. Τρία σημεία θα ήθελα να τονίσω. Είναι σημαντικό, θεωρώ, η ρύθμιση αυτή Ε, είναι σημαντικό το γεγονό ότι η ρύθμιση αυτή ε, προβλέπει μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Δεν τα μειώνει όμως τα απόβλητα αυτά, γι' αυτό είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή για τις συνέπειες ε, των αγορών του. Είναι σημαντική μετά και πέρα από την ευθύνη του παραγωγού και η ευθύνη του καταναλωτή. Σύμφωνα με την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, θα πρέπει να υπάρχει και η αρχή της επιβάρυνσης του παραγωγού και του καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε επίσης ε, την επαναχρησιμοποίηση σπάνιων πρώτων υλών. Εμείς ο στόχο, στην τελική ανάλυση, έχουμε το 100% της επαναχρησιμοποίησης και αυτό θα πρέπει να προβλέπεται και στη φάση του σχεδιασμού του κάθε προϊόντος γιατί τελικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία θα προβλέπει το τέλος της ζωής κάθε συσκευής. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη αυτό κατά τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων και σε ό,τι αφορά και την προευθύνη του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρδίνη. Θα είμαι πολύ σύντομη πρόεδρε, τα περισσότερα υπόθηκαν. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα πολύ σημαντικό, αλλά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περιπεπλεγμένη. Γι' αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ με τρία σημεία κρίνω πως ε, το να θεωρήσουμε ότι η παραγωγή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την χρηματοδότηση της όλης ε, διαδρομής ε, από την αγορά μέχρι το τελική χρήση, τελική χρήση του, της συσκευής δεν είναι σωστό εξάλλου. Θεωρώ ότι αυτό δεν που επηρεάζει ούτε το ζήτημα των ε, παράνομων εξαγωγών, ούτε της παράνομης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επηρεάζει επίσης και την ευαισθησία και ευαισθητοποίηση των πολιτών μας. Είναι βασικό βασικός στόχος αυτός, θα θέλουμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα επί συγκεκριμένων κατηγοριών που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες. Πιστεύω επίσης ότι χρειάζεται να αναλάβουν τα κράτη-μέλη την ε, το στόχο της επίτευξης ε, ενός υψηλού ποσοστού. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καταλήτως τρόπος για να υπάρξει η μεγάλη συμμετοχή των εμπλεκομένων και τρίτων που θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι πως εάν θελήσουμε να αναθεωρήσουμε το πεδίο εφαρμογής τότε θα πρέπει να επαληθεύσουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει οι συνέπειε αυτής τη οδηγία. Δεν συμφωνώ διόλου με τον αρνητικό πίνακα των προϊόντων να πούμε ότι εκτό από αυτά τα προϊόντα τα υπόλοιπα θα πρέπει να διευρυνθούν περαιτέρω. Αυτά ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, έκθεση του που βρίσκω ιδιαίτερα σημαντική. Μερικές σύντομες ε, σκέψεις. Ε, μετά από συζητήσεις που είχαμε τους παραγωγούς διαπίστωσα το ενδιαφέρον τους σχετικά με την ανάληψη της πλήρους ευθύνης για το προϊόν. Αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τι εννοώ υπάρχουν κάποιες παράλληλες γραμμές που όμως ε, διακινδυνεύουν να ανακτήσουν το πιο πολύτιμο τμήμα του αποβλήτου και να αφήσουν το υπόλοιπο στο τύχη του. Θεωρώ λοιπόν πως οι παραγωγοί θα πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι και αυτό έχει πρώτη στη σημασία. Επιθυμώ επίσης να πω πως συμφωνώ σε ό,τι αφορά τα μικρές συσκευές όπως λαμπτήρες ή οτιδήποτε άλλο αυτά θα πρέπει να συλλέγονται με την συμμετοχή του λιανοπολιτή. Να τονίσω επίσης την ε, διαφορετική ρύθμιση που ζήτησα για τα ηλιακά κάτωπτρα διότι δεν πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και οποία είναι εγγυημένα για περίοδους ε, τουλάχιστον 20 ετών και άνω και άρα μπορούν στην ουσία αυτόματα να αποκτούν το ενδιαφέρον των παραγωγών για να τα ανακτούν και να τα ανακυκλώνουν. Πρόκειται για έναν κλάδο που θα πρέπει να ρυθμιστεί ιδιαίτερα και ειδικά. Ευχαριστώ. Φρονσουάς Γκροστέντ λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε για την ποιητή της έκθεσης Φλόρενς. Υπάρχει κάποια δυσκολία σε ό,τι φορά τον ορισμό του παραγωγού. Ο παραγωγός θα πρέπει να καταγράφει το προϊόν του. Ε, στην πραγματικότητα πρόκειται για απόβλητο, διότι το προϊόν μετά από τη χρήση θα καταστεί απόβλητο και ο παραγωγός θα πρέπει να ε, γράφεται στο κράτος μέλος στο, στο οποίο το προϊόν του θα καταστεί απόβλητο διαφορετικά δεδομένου ότι υπάρχει ελευθερία και κυκλοφορία των προϊόντων στην ιστορική αγορά, ε, επιτρέπουμε ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία των αποβλήτων. Αυτό όμως το θέλουμε να το απαγορεύσουμε. Άρα ο ορισμός του παραγωγού θα πρέπει να είναι εθνικός. εθνικός. Διαφορετικά θα υπάρξει ο κίνδυνος ε, ενός τουρισμού αποβλήτων. Η πρόταση λοιπόν της ε, Κομισιόν είναι ευαίσθητη σε σημείο αυτό, είναι τρωτή λοιπόν. Έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες ε, πάνω στο ζήτημα αυτό τώρα για το θέμα του περιβάλλοντος ή την ε, οικοσυμβολή θα πρέπει να αναφέρεται αυτή η επισήμανση. Τώρα για το σύστημα της ανάκτησης και της, της συλλογή μάλλον θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για όλα τα σημεία ε, τα οποία μπορεί να ε, μεταφέρει το απόβλητο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσοστό των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που συλλέγονται προς ε, επαναχρησιμοποίηση. Αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση που ακολουθεί, το βαθμό 8, θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες συγκεκριμένε ε, ε απαιτήσει ε, όπως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ηλιακά κάτωτρα. Κύριο Σόνικ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και τον εισηγητή που έλαβε υπόψη του το αίτημά μας ε, σχετικά με την ε, συλλογή στις επιμέρους χώρες και είχα κατά νου τις λιγότερο αντιμένες χώρες. Εάν ε, θέλουμε λοιπόν το κείμενο αυτό να στεφθεί από επιτυχία θα πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στα επιμέρους κράτη μιλούσαμε για εισαγωγές, εξαγωγές και επιθυμώ να πιστήσω την προσοχή σας σχετικά με τις απάτες. Παραδείγματος χάρη η πλαστογράφηση κάποιων ε, αποδείξεων, ε, κάποιων τιμολογίων. Δημιουργούνται, συστήνονται εταιρείε ε, μόνο και μόνο για να συμπληρώνουν αυτά τα τιμολόγια τα οποία είναι πλαστά και διαρωτώ με πώς θα μπορούσε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν κατά πόσο η Κομισιόν έχει μια πρόταση, κάτι το οποίο θα επέτρεπε τα κράτη-μέλη και θα υπορρένουν μάλλον τα κράτη-μέλη να ελέγχουν παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει ένα νομικό κενό μερικές φορές, άλλες φορές υπάρχει μια ανοχή. Εδώ έχω ένα έγγραφο πολλών σελίδων το οποίο περιγράφει την ε, λειτουργία αυτού του συστήματος ε, στην Πολωνία. Το ε, κείμενο αυτό αφορά την συλλογή των συσκευών στην Πολωνία και η κατάσταση αυτή πραγματικά με εντυπωσιάζει και με φοβίζει συνάμα. Δεν ξέρω κατά πόσον οι μεγάλες μας φιλοδοξίες δεν θα παραμείνουν νεκρό γράμμα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να μεταφραστεί στην πράξη αυτή η βούλησή μας. Η Κομισιόν θα πρέπει να βουλέψει μηχανισμούς ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες 27 και 28 γιατί να μην αναλάβει ο παραγωγός, ο ε, το κόστος. Εάν βγάλουμε δηλαδή έξω ένα συγκεκριμένο κλάδο, όπως αναφέρεται στην τροπολογία 9, τότε αυτή η αιτιολόγηση εδώ είναι κάπως περίεργο. Αναφέρεται δηλαδή ότι μέχρι το 2014 θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι το 85% των φωτοβολταϊκών μονάδων έχει ανακυκλωθεί. Ο Βιτόριο Πρόντι ε, είπε ε, πως ε, έχουν διάρκεια ζωής 20 με 25 έτη αυτές οι μονάδες. Άρα λοιπόν μέσα στα, σε αυτές τα, τα επόμενα χρόνια δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν στοιχεία ίσως από το 2034 και μετά δεν ξέρω. Δηλαδή η διατύπωση εδώ είναι κάπως λανθασμένη. Η κυρία Καντίνα Φάσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τώρα το λόγο και θα έχουμε στο τέλος και Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπής. Ε, διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον σε όλε αυτέ αυτές τις οι διαφορετικές απόψεις οι οποίες εκφράζονται ε, απηχούν και τη μεγάλη σημασία αυτής της ε, νομοθετικής ε, πράξης αλλά μας δίνει και μια εντύπωση για τις προσπάθειες που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των εργασιών του για αυτό το νομοθέτημα. Στο σύνολό τους θεωρούμε πως αυτές οι τροπολογίες εκφράζουν υποστήριξη για τα κύρια στοιχεία της πρότασης Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση τη ιατρικής οδηγία και αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Δηλαδή η ε, ε, λάτωση αν θέλετε της ε, εκτεταμένης, του εκτεταμένου αν θέλετε, τρόπου χειρισμού μέχρι στιγμής αυτών των συσκευών, η αύξηση του ελέγχου και ταυτόχρονα και η πρόληψη των, α, της μεταφοράς αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδικότερα σε χώρες στις οποίες η επεξεργασία αυτών των αποβλήτων θα γίνει με τρόπο ο οποίος δεν είναι αντίστοιχος με αυτό στην Ευρώπη. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο τονίστηκε επανειλημμένα σήμερα ήταν η ανάγκη για ένα φιλόδοξο στόχο συλλογή των συσκευών, στόχο τον οποίο καλωσορίζουμε, αλλά ε, και ύπαρξη ενό στόχου ο οποίο θα ανταποκρίνεται στη διαφορετική πραγματικότητα των εκάστοτε κρατών μελών. Θεωρούμε πω είναι ένα σημαντικό τρόπο για την αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση για να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτόν τον στόχο, υπήρξαν μια σειρά από σχόλια. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο του στόχου, καταρχήν, δηλαδή το 65% όπω αυτό προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε πω το 85% των παραγόμενων αποβλήτων είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που εμείς προτείνουμε, δηλαδή βρίσκεται κοντά στο 65% των αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε, αν θέλετε, μια μετατόπιση από το που βασιζόμαστε στο ποσοστό, αλλά θα χρειαστεί να συζητήσουμε εδώ μια εναρμονισμένη μεθοδολογία ως προς την παρακολούθηση, την εποπτεία δηλαδή της στήριξης αυτού του στόχου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό και η δική μας εμπειρία στο πλαίσιο της εφαρμογής ε, νομοθεσίας μας δείχνει ότι θα χρειαστούμε κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή θα χρειαστούμε και μια αντίστοιχη εντολή επιτροπολογίας ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες, συγκεκριμένοι κανόνες, εναρμονισμένοι κανόνες ως προς το πώς θα παρακολουθείτε η τήρηση αυτού του ποσοστού. Μετά τέθηκε το ζήτημα διαφοροποιημένων στόχων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά μικροηλεκτρονικές συσκευές δηλαδή ξεχωριστού στόχου. Ο στόχο ω τέτοιο, το ποσοστό δηλαδή είναι ε, κάτι το θεμελιώδε μέσα στην πρόταση και θα πρέπει να διασφαλιστεί πω ε, η φιλοδοξία μα εδώ δεν μειώνεται. Ταυτόχρονα όμω θεωρούμε πω η διαφορετική πραγματικότητα που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει και εκείνη να ληφθεί υπόψη ε, κατά την διατύπωση, κατά την εκπόνηση του αντίστοιχου στόχου. Και αυτό ισχύει ειδικότερα σε ό,τι αφορά κάποιες μικρές, κάποια μικρά κομμάτια της αγοράς. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, ε, τον στόχο, ε, ε, ένα συγκεκριμένο στόχο σε ό,τι αφορά τα, τις συσκευές και τον εξοπλισμό ψήξης και θέμας, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε στο 2012, δηλαδή να έχουμε μια έκθεση όπου θα εξετάζουμε ακριβώς την θέσπιση ενός ξεχωριστού στόχου. Γιατί μιλάμε ε, βέβαια για συσκευές εδώ οι οποίες ούτως ή άλλως δεν αποτελούν το κύριο σημείο ανησυχία ε, των περισσότερων ε, μελών της Επιτροπής εδώ και του Κοινοβουλίου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε και λαμπτήρες που έχουν ράδιο ή οτιδήποτε άλλο το οποίο ενδέχεται να χρειάζεται να τύχει ξεχωριστής μεταχείριση στο πλαίσιο του στόχου. Επίσης, υπογραμμίζουμε τις τροπολογίες εκείνες και τις σημασίες τους που αναφέρονται στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στο ίδιο πλαίσιο κάνουν λόγο για ε, την αποφυγή ε, περί του διοικητικού φόρτου εργασίας ειδικότερα τροπολογίες εκείνε, οι οποίες στήγουν το άρθρο 16 σε ό,τι αφορά ε, την καταχώρηση, την παροχή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων, όπως και οι τροπολογίες που αφορούν τον ορισμό του κατασκευαστή. Θεωρούμε πως τα άρθρα 3 και 16 είναι πάρα πολύ σημαντικά για την, να επιτύχουμε την ε, μείωση του ε, διοικητικού άρθρους. Ε, ήταν ε, κάτι πολύ σημαντικό που ελήφθη υπόψη στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας και νομίζουμε πως αυτό το στόχο το συμμερίζονται και πάρα πολλοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν οι τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν ερμηνεύονται από εμά ως τροπολογίες που κατευθύνονται προς τον ίδιο στόχο. Αυτό λοιπόν το νέο νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να θέσει ένα τέλος στις ε, μη εναρμονισμένες ε, μεθοδολογίες και στους τρόπους εργασίας των κρατών Ταυτόχρονα θα πρέπει να μην επιβάλλεται πλέον ε, ε, πολλαπλή αν θέλετε πληρωμή για τη μεταχείριση ενός και μόνο προϊόντος και τέλος θα πρέπει να λάβει τέλος η πρακτική του να πρέπει να υπάρχει μια νόμιμη έδρα για το κάθε ξεχωριστό προϊόν. Ε, που διατίθεται εκεί. Κλείνω εδώ, ε, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ ξανά για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω από τον κύριο Φλόρεντς ε, να περιοριστεί στα τρία λεπτά, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο για την έκθεση Evans. Ναι, ευχαρίστω να το κάνω. Θα ήθελα να πω στους συναντέλφους από τη, χώρα μας, από τη χώρα μου που θέλουν το 85% ως ποσοστό επαναχρησιμοποίησης, ενώ στις ε, άλλες χώρες, ε, στις πιο αποτελεσματικές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κόσμος διαμαρτύρεται και για το 65%. Να τονίσουμε λοιπόν πόσο αντικρουόμενα είναι τα συμφέροντα με το 65%. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Να δούμε αν θα το καταφέρουμε κιόλα. Το πολύ σημαντικό είναι η τυποποίηση κάποιων συγκεκριμένων ε, ζητημάτων. Όπως για παράδειγμα οι οδηγίες πλαίσιο, οι οποίες όμως ε, εφαρμόζονται Ξέρω και παράδειγμα ότι στην Αυστρία και στις σκανδιναβικές ε, χώρες είναι πάρα πολύ σωστός ορισμός των σημείων συλλογής, αλλά δεν ισχύει αυτό σε χώρες γειτονικέ της Αυστρίας και γι' αυτό έχουμε τέτοιες επιστροφές, γιατί θα πρέπει να πληρούνται πάντα τα συγκεκριμένα κριτήρια για να υπολογίζουμε σωστά τις ποσοστώσεις, τα ποσοστά. Φυσικά και εγώ θέλω να υπάρχουν πολύ πιο υψηλά ποσοστά, αλλά δυστυχώ κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλίστες και το ερώτημα του ποιες θα είναι οι παράμετροι που θα εφαρμοστούν. Put on the market ή σε ό,τι αφορά την θέση στην ροή. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τα ηλιακά πάνελ. Νομίζω ότι η βιομηχανία ο κλάδος είναι σε θέση να αποδείξει ότι και χωρίς ευρωπαϊκή ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει. Το έχουν ήδη αποδείξει άλλωστε. Και έχουμε τρία χρόνια στη διάθεσή μας ε, για να το πιστοποιήσουμε αυτό, να το τεκμηριώσουμε και αν δεν τεκμηριωθεί θα υπαχθούν αυτόματα μετά από τρία έτη στην νομοθεσία αυτή. Αυτό αποτελεί απλά μία πρόταση την οποία θα υπέβαλα. Δεν πρόκειται να υπεραμυθώ αυτής. Ο Κρις ζητάει να ορίζονται με σαφήνεια οι φορείς συλλογής Μακρίστ. Είναι τώρα αυτό φιλελεύθερη πρόταση. Το αντίθετο μου φαίνεται και οι Ιταλοί συνάδελφοι λένε να ορίσουμε σχετικά κριτήρια. Εγώ είμαι υπέρ του να οριστούν κριτήρια. Θέλω να υπάρχει αυτό το φιλελεύθερο στοιχείο. Θεωρώ ότι είναι καλή στο σημείο αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό την άλλαξα. Γιατί δεν διστάζω, ξέρετε, να επιτεθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όταν τα έχει πάει καλά δεν υπάρχει λόγος, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ να ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος, στις 4 Μαΐου στην Επιτροπή για την έκθεση αυτή και τον Ιούνιο ελπίζουμε πριν από τις θερινές διακοπές να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και να περάσουμε σε ένα παρόμοιο θέμα στην έκθεση της G11 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Να δώσω κατευθείαν το λόγο στην εισηγήτρια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά σας παρακαλώ μην υπερβείτε τα πέντε λεπτά για να διευκολύνετε και τους συναδέλφους μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπερβώ τα πέντε λεπτά γιατί πολλοί συνάδελφοι τόνισαν και στην προηγούμενη συζήτηση την ανάγκη να κυκλώνονται κάποια υλικά, κάποιες πρώτες ε, ε, ύλες να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες στην έκθεσή μου. 339 στον αριθμό. Δεν έχουν μεταφραστεί όλες τους ε, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, όχι ακόμα. Το πλήρες ε, κείμενο στα αγγλικά το έλαβα και εγώ μόλις σήμερα. Θα χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολύ χρονικό διάστημα για να εξετάσουμε το περιεχόμενο και να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Και φυσικά να δούμε και πού είναι οι διαφορές μας. Να σας δώσω λοιπόν μία αρχική εντύπωση σήμερα. Σκοπός μου όμως είναι να το συζητήσω αυτό με τους συναδέλφους, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες και να σημειώσουμε και πρόοδο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την έκταση του προβλήματος των αποβλήτων που αντιμετωπίζουμε, το σύνολο που εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το 2020 σε 12 εκατομμύρια τόνους και σκοπός ήταν να αποτραπεί η δημιουργία αποβλήτων. Αυτό το πετύχαμε και θέσαμε παγκόσμια πρότυπα. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ευθύνη σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση αυτή της νομοθεσίας αυτής και υποστηρίζω τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι να καταστεί πιο ε, κατανοητή και πιο εφαρμόσιμη αυτή η νομοθεσία. Ξέρουμε ότι πολλές εταιρείε έχουν υπερβεί ήδη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και έχουν καταργήσει τις επιβλαντές φλόγας, τα λαγονούχα επιβλητικά φλόγας. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να επικεντρωθώ στα βασικά θέματα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή καταρχάς. Θεωρώ ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτονται. Γιατί αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο να υπάρχει νομική βεβαιότητα. Και αυτό αποτελεί και στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τροπολογίε δείχνουν ότι πολλές ομάδες ε, υποστηρίζουν αυτή την αρχή, αλλά πολλές ομάδες έχουν κάνει τροπολογίε για εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, μέσα μεταφοράς, μεγάλες εγκαταστάσεις και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό και να το συζητήσουμε. Καλώς ορίζω και δέχομαι την ε, τροπολογία 148 των σοσιαλιστών για την ευθύνη όλων των φορέων για τη μείωση της έκθεσης ε, στον καταναλωτή και στο περιβάλλον και οι απόψεις είναι αντικρουόμενες ε, σε ό,τι αφορά τα ελιακά κάτωπτρα, κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχει μια πρόταση να καταργηθούν τα προϊόντα που περιέχουν κάδμιο και να εξαιρεθούν στο σύνολό τους οι ανανεώσιμες. Ε. Εγώ προτείνω προσωρινή εξαίρεση ανάλογα και με τα απορίσματα των ε, ερευνών. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα τα υλικά των εκτυπωτών. Ένα δεύτερο θέμα είναι η σχέση με το REACH. Όπως ανέφερα στο παρελθόν, υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν μπορεί το ΡΙΤΣ να αντικαταστήσει το την νομοθεσία αυτή, η οποία καταρτίστηκε για συγκεκριμένα προβλήματα του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ορίζει ότι τα δύο νομοθετήματα είναι συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση των δύο, συνένωση των δύο νομοθετημάτων και θεωρώ ότι η ΡΟΣ έχει αποδειχτεί επιτυχής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ξεχωριστή μεθοδολογία. Και πάλι, πολλές τροπολογίες έχουν υποβληθεί για το θέμα αυτό. Εγώ πρότεινα στην έκθεση να καταργηθούν μετά από τρία έτη μετά την επαναδιατύπωση και τη θέση της έσχη των αλλαγονούχων επιβραδυτικών φλόγα και των PVC και συμπεριλαμβάνω συγκεκριμένη αναφορά του Ινστιτούτου του Ιδρύματος ΕΚΟ που διεξήγει σχετική έρευνα και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν τεθεί τροπολογίες για το παράρτημα υπαριθμών 3. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις έρευνες που έχουν γίνει στα παρελθόν. Αλλά όπως είπα, οι μεγάλες εταιρείε προηγούνται ήδη των προτύπων αυτών. Άρα θεωρώ ότι το επόμενο λογικό βήμα είναι να επεκταθούν οι περιορισμοί. Διάφορες προτάσεις επίσης έγιναν για την μεθοδολογία που ασφαλώς αποτελεί κεντρικό σημείο κλειδί και η διαδικασία για τη χορήγηση εξαιρέσεων ασφαλώς αποτελεί ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Άρα θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε με τον γενικότερο στόχο ότι θα πρέπει να καταστεί πιο αποδοτική η νομοθεσία αυτή και όπως είπα και στην αρχή αντιμετωπίζουμε την πιο ταχαίως αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων και θα πρέπει λοιπόν ανάλογα να την αντιμετωπίσουμε. Θα έρθω σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές για να συζητήσουμε ξεχωριστά τα θέματα αυτά και να καταλήξουμε όπου είναι δυνατόν στη συμφωνία. Thank you Ευχαριστούμε την κυρία Evans και να περάσουμε στους, ε, στους ε, σε όσους έχουν ζητήσει το λόγο 10 ομιλητές, να περιοριστούμε στα δύο λεπτά. Ο κύριος Σόνικ. Λοιπόν, Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ πρότεινα μία δομή η οποία μπορεί να βάλει τάξη στα πράγματα και θα σας ε, παρουσιάσω αυτή την λύση. Το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία ε, θα πρέπει να υπάρξει, να συμπεριληφθεί όλο ο ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θέσει τέρμα στα προβλήματα ερμηνεία ε, και την έλλειψη σαφήνεια. Δεύτερον, προτείνω έναν, ένα μητρό, έναν κατάλογο με όλε τι εξαιρέσει θα αφορούν, αφορούν ομάδες ε, συσκευών συγκεκριμένη ε, χρήση σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόβλητες στις περιπτώσεις σε αυτές τις, ε, τις Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και θα υπάρχει και μια ε, ερμηνεία. Θεωρώ ότι η οδηγία αυτή έχει ανάγκη από σαφείς ορισμούς και περιορισμό των ουσιών, θα πρέπει να πούμε ποια είναι τα κριτήρια για την εξέταση κάθε ουσίας σε συγκεκριμένε φάσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε εδώ τη διαδικασία του Ρίτς. Η απαγόρευση μιας συγκεκριμένη ουσίας θα πρέπει να ε, γίνεται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και αποτελέσματα ότι η ουσία αυτή είναι επικίνδυνη και ο κίνδυνος τον οποίο παρουσιάζει δεν μπορεί να περιοριστεί. Αυτές οι εξαιρέσεις λοιπόν που προτείνω, ε, προτείνω να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η ε, ομάδα Α με τέσσερα έτη ως περίοδο αναθεώρησης, εάν η μείωση μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατή και σκόπιμη, και η ομάδα Β με προϊόντα που χρησιμοποιούν τις, ε, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά απαγορευμένων ουσιών και που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί αυτή η επικίνδυνη πλαβερή ουσία και εδώ η περίοδος αναθεώρησης θα είναι δεκαετής ε, διάρκειας. Δύο κατηγορίες λοιπόν εξαιρέσεων. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά επόμενος αγορητής, ε, αγορήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στην πρόταση της Χίδριας προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες να καρελεθούν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες θα μπορέσουν να υποστηριχθούν από ε, την ψηφία των μελών της Επιτροπής μας και πως ε, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά, να δει το, και αυτό να το δείξουμε, να μιλήσουμε για ουσίες που θέλουμε να καταργήσουμε και να είμαστε πραγματικά πιστικοί με τις εργασίες μας. Αν είμαστε όλοι λοιπόν πεπισμένοι περί αυτού, τότε οι τροπολογίες μας θα είναι αποτελεσματικές και η επιτυχία της οδηγίας θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις τροπολογίες αυτές. Όλα αυτά πράγματι θα λειτουργήσουν ελπίζω με τους ομιλητές. Ο κύριος Δέβης. Ε, σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, ναι, ε, ελπίζω πως ε, θα υπάρξουν, ε, θα, θα μπορέσει η συγκήτρια να πετύχει κάποια πράγματα, αλλά όχι με εμά. Κάποιες άλλες συμβαστικές τροπολογίες θα είναι πιο δύσκολες. Από τους πράσινους συναδέλφους. Και γνωρίζω πως συνάδελφος θέλει πάντα να τονίζει πως είναι ε, σε περισσότερο εθνική κατεύθυνση και όχι πράσινη. Εν πάση περιπτώσει, ε, συμφωνούμε με την κατεύθυνση στην οποία ακολουθεί εδώ η συγκήτρια, συμφωνούμε με το πεδίο εφαρμογή, αλλά χρειαζόμαστε εδώ μια σειρά από σαφεί εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογή αυτό. Ε, θα πρέπει να έχουμε εδώ μια όθηση που να δείχνει ότι θέλουμε ε, να έχουμε εδώ αντικατάσταση περισσότερο βλαβερό με λιγότερο βλαβερέ ε, ουσίες, ε, ε, όχι όμως πλήρη κατάργηση χωρίς να έχουμε συγκεκριμένες αξιολογήσεις εδώ, εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο και θα πράγματι και συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κανονισμό και να διασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα και ένα κοινό στόχο. Άρα λοιπόν αναμενούμε με ενδιαφέρον τι επόμενε τέσσερι εβδομάδε, ούτω ώστε να πετύχουμε να κάνουμε κάτι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γκένι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πεδίο εφαρμογή. Δεν θεωρώ πω ε, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να επισέλθουμε σε εκτενεί εντοσυζητήσει. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να διαπραγματευτεί το παιδί εφαρμογή με τον τρόπο που προτείνεται. Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι πολύ ε, επιπλαβέ. Ε, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τι εξαιρέσει. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή πώ με ένα πρόβλημα θα επιληθεί ένα άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν πρωτού προβούμε σε τέτοιες ε, εκτεταμένες αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, τροποποιήσεις που προτείνονται για το παράδειγμα, ε, έχουμε εδώ κάποιες προτινόμενες απαγορεύσεις ορισμένων ουσιών, χωρίς όμως να επιλύονται εδώ ε, κάποιες οργανικές δηλαδή ενώσεις και χλωρίου και ευρωμίου σε ό,τι αφορά τα επιβερδυτικά φλόγα και το ε, PVC δεν υπάρχει εδώ μια αιτιολόγηση γιατί πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο η απαγόρευση Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι επανειλημμένα έχουν απευθυνθεί επιχειρήσεις σε εμάς ότι ε, γίνονται κάποιες αλλαγές και πράγματι γίνονται αλλαγές στις ε, διάφορες κατηγορίες αλλά ε, δεν, δεν νομίζω πως στην πλειοψηφία αυτών των κατηγοριών γίνονται έτσι αυτόματα όλες αυτές οι αλλαγές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, προσεκτικά αυτές τις αλλαγές και να δούμε τι ακριβώς θα ε, ποιο θα είναι ο αντίκτυπο τέτοιων απαγορεύσεων σε ό,τι αφορά τα υποκατάστατα. Δεν έχουν αξιολογηθεί τα χαρακτηριστικά του ε, πλήρω ακόμα. Ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιε ωφέλειε ε, για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν 75 διαφορετικά υποκατάστατα, οπότε θα πρέπει να τα εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα. Ε, επίσης υπάρχει και το ζήτημα των μη ρυθμιζόμενων, δηλαδή των μη ελεγχόμενων αποβλήτων, ο Καλαγιάννης Φρόνες ανέφερε το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα των εξαγωγών αποβλήτων που δεν ελέγχονται και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και όχι στην απαγόρευση των ουσιών. Επόμενο ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την G. Ε, Levans την εισηγήτρια, για μια πολύ καλή πρόταση γνωμοδότηση, η οποία βελτιώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια σειρά από σημαντικά σημεία. Ωστόσο, δεν συμπαρατάσσομαι με την διάταξη για την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογή των φωτοβολταϊκών μονάδων που περιέχουν κάδμιο. Ε, νομίζω πως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια ε, η της κατασκευής αλλά Υπάρχουν και ταυτόχρονα υποκατάστατα που ήδη εφαρμόζονται από διάφορους κατασκευαστές, αλλά λοιπόν μέχρι το 2015 θεωρώ πως θα είναι δυνατή ε, ή πάυση, διακοπή δηλαδή της κατασκευής τέτοιων μονάδων. Επίσης ε, θέλουμε περισσότερες, ε, περισσότερους περιορισμούς σε ό,τι αφορά ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Αναφέρονται πολλές ουσίες εδώ, αλλά περιλαμβάνονται αυτές στο παράρτημα 3. Εμείς λοιπόν ζητούμε με τη δική μας τροπολογία οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες να περιληφθούν στο παράρτημα 4. Δηλαδή να περιληφθούν στις απαγορευμένες ουσίες, καθώς η, χρήση τέτοιων ουσιών έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για, τον, για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, πράγμα το οποίο είναι είναι ανεύθυνα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα βρωμιούχα ε, επιβραδυτικά βλόγος ε, μπορούν να βρεθούν σε ό,τι αφορά δηλαδή πολύματά τους μέχρι και στο μετρικό γάλα. υπάρχουν και περισσότερες ε, ουσίες. Στο παράδειγμα 4 ωστόσο δεν υπάρχουν κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας δείχνουν τέτοιου είδους να είναι ενδεχομένως να είναι προβληματικά. Επίση, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην τοπολογία μου 313, η οποία αφορά το παράδειγμα 4 και τι επιτροπένε ανώτατε συγκεντρώσει. Εδώ αναφέρονται λοιπόν ε, οργανικές ενώσεις φλόρου και άλλα δρομούχα επιβραδυτικά φλόγας. Ε, στα γερμανικά λοιπόν υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα μετάφρασης γιατί στα αγγλικά αναφέρονται other undominated και ούτω δυτικά φλόγες. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα αυτή η διάκριση που έγινε από την ε, εισηγήτρια ανάμεσα στο Ρίτσουδιο και το Ρώσο. Το ένα είναι ποσοτικό, το άλλο ποιοτικό. Τα λέω όλα αυτά πρώτα απ' όλα διότι το θέμα της ε, των υποκατάστασης ε, ορίζονται σε πολλές περιπτώσεις. Ε, υπάρχει το θέμα των ε, υπολογιστών που λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ασήμι και όχι μόλιδο. Κοιτάξτε, ο καταναλωτής δεν τρώει τον υπολογιστή, δεν είναι βρόσιμος. Λοιπόν, και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις θέσεις του Σόνι να κάνουμε μια ταξινόμηση. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφής αυτή η ταξινόμηση, αυτή η κατηγοριοποίηση. Επανειλημμένα λοιπόν έχουμε ε, πάρει αποφάσεις κατά του ιστορικής και πολιτικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να κλείσουμε λοιπόν όλα τα μουσεία που έχουν ε, αρχαιολογικά αντικείμενα μέσα. Σε πολλές πτυχές λοιπόν χρειαζόμαστε να έχουμε σαφή παραδείγματα. Ένα ζήτημα είναι αυτό το θέμα των ιστορικών αντικειμένων, των πολιτικών στοιχείων, τα οποία χρειάζεται και να τα ρυθμίσουμε, να τα λάβουμε υπόψη για να, για να φέρουμε μάλιστα σε κάποια μουσικά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούν και στις εκκλησίες μας και στα θέατρά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ιστορική πολιτική κληρονομιά και θα πρέπει η Κομισιό να το λάβει υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ναι, του υπολογιστέ έφερε το στρώμα. Το μάθαμε και αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αναφερθώ στην ανάγκη συντονισμού με την οδηγία REACH. δεν πρόκειται για συγχώνευση αλλά για εναρμόνιση. Περιφορά τις διαδικασίες ε, ελέγχου που αφορούν στο ρίτσο θα πρέπει να εφαρμοστούν και στις οδηγίες και στις ουσίες αυτού της, του οργανισμού. και θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα είδος μιλφέγγι το οποίο θα καταστεί ε, αχώνευτο από τον οργανισμό. Νομίζω η τροπολογία της ε, γροστέτ που αφορά το σημείο 1,7 είναι το κατάλληλο και ζητάει την απόσταση του ΠΔΣΑ από τους ουσίες που θα πρέπει να απαγορευτούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Φωνσός ε, Γκροστέτ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ για το πεδίο εφαρμογή Είτε ζητάμε πολλές εξαιρεσει και τότε θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Τροπή που δεν θα ξέρει πώς θα αποφανθεί επί του θέματος το αντίστροφο θα έχουμε τόσε πολλέ εξαιρέσεις που η νομοθεσία θα καταστεί αναποτελεσματική, κάτι το οποίο θα είναι λυπηρό. Θα πρέπει να διατηρήσουμε και την αερογωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και εδώ θα επανέλθω στα όσα υπόθηκαν, θα πρέπει να αποφύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας καλός συντονισμός και διάρθρωση με το REACH που θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από την οδηγία αυτή. Λοιπόν, αποκλείσουμε για επειδή εφαρμογή οδηγία ε, κάποιον εξοπλισμό που αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη, παραδείγματο χάρη κάποια, ε, κάποια ιατρικά βοηθήματα όπω peacemaker κλπ. Μιλήσαμε επίση και για το PVC, δεν επανέρχομαι και επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε εξαιρέσει σε ό,τι αφορά τα ηλιακά κάτωπτρα. Υπήρξε ένα λάθο μετάφραση ε, στα αγγλικά όπου μιλάμε για αποκλεισμό, συγγνώμη, μιλήσαμε για εξαίρεση, ε, μιλάει για εξαίρεση, αλλά εγώ θέλω να πούμε για αποκλεισμό. Οι δύο όροι είναι συγγενικοί, αλλά δεν αφορούν στο ίδιο πράγμα. Κυρία Καρδίνη, το λόγο. Θα είμαι σύντομη και θα αναφερθώ στο πεδίο εφαρμογής με τα όσα ακούσαμε κατέστη προφανές ότι το να συμπεριληφθούν όλα τα, όλες τις συσκευές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσουμε τα θέματα ερμηνείας σε ό,τι φορά το πεδίο εφαρμογή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες, σαφείς, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να διευρύνουμε σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές εάν δεν αξιολογηθούν καλύτερα οι συνέπειες δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά και μάλλον θα υπάρξουν και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Θεωρώ ότι το κείμενο της Κομισιόν Ερωταποκρίσεων του Μαΐου του 2005 είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για το θέμα του πεδίου σας. Σταματώ εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να... να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρία λεπτά, αν μπορείτε να περιοριστείτε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κι εμείς αρκετά γρήγοροι να υποθυμίσουμε ότι αυτή η αναδιατύπωση περιλαμβάνει την εξέταση μιας νομοθεσίας η οποία είναι ακόμα σχετικά πρόσφατη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό είχε να εξυγχρονίσει και να απλοποιήσει μια τέτοια νομοθεσία η οποία έχει αντίκτυπο σε πολλούς οικονομικούς φορείς. Αυτό να το έχουμε υπόψη σε ό,τι αφορά και την υποβολή των τροπολογιών και τροποποίησεων ε, του κειμένου της οδηγίας. Κάποια θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ε, αναδιατύπωση των δύο αυτών οδηγιών για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα θέματα τα οποία προέκυψαν σε ό,τι αφορά τις δύο οδηγίες. Το πεδίο εφαρμογής και η επέκτασή του δεν περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν περιλήφθηκε στην έκταση αντικτύπου. Δεν υποστηρίζουμε λοιπόν την τροποποίηση σημαντικών τμήματων των οδηγιών χωρίς σωστή μελέτη αντικτύπου. Ίσως να χρειαστούν κάποιες νέες εξαιρέσεις και αυτό το επιβεβαίωσαν και οι συμβολές σας σε ό,τι αφορά η μελλοντική ερμηνεία των ε, τροπολογιών αυτών ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγάλη ασάφεια σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νέες ουσίες, τις νέες ομάδες ουσίες οι οποίες ε, προτείνονται, προτείνονται να περιοριστούν με επιχειρήματα κάποιων ερευνών. Δεν θεωρούμε ότι τα πορίσματα της έρευνας επαρκούν για τον περιορισμό των ουσιών αυτών. Δεν θεωρούμε ότι δικαιολογούν τέτοιες προτάσεις. Θεωρούμε λοιπόν και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι για να γίνουν περιορισμοί τέτοιοι και εξαιρέσεις τέτοιοι, τέτοιες θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα επιστημονικά πορίσματα και Επίσης, ε, μελέτες αντικτύπου για την ενδεχόμενη συνέπεια των απαγορεύσεων αυτών. Τέλος, να σημειώσω ότι με χαρά μου παρατηρήσω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που διευκρινίζουν τους ορισμούς που προτείνονται για τις διαδικασίες εξαίρεσης, για τη μεθολογία περιορισμών που ουσιαστικά υποστηρίζουν τους στόχους της αναδιατύπωσης αυτής και ευχαρίστως να τη συζητήσουμε περαιτέρω. Για να ολοκληρώσουμε τώρα, να ολοκληρώσω τα σχόλια αυτά, να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει να εξεύρουμε μια ισορροπία σε αυτή την αναδιατύπωση για να διατηρήσουμε τα όσα έχουν λειτουργήσει σωστά ως τώρα και παράλληλα φυσικά να εξυγχρονίσουμε το νομοθέτημα αυτό για να αποτελέσει μια σωστή βάση για ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας ή των ε, ομάδων των ουσιών. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε δύο λεπτά στην εισηγήτρια αν κυρίως ό,τι αφορά το θέμα της μελέτης αντικτύπου για την επαγόρευση επικίνδυνων ουσιών. Δεν ήταν σαφές στην επεξήγησή σας, γιατί αναφέρεται σε ένα σημείο ότι πρόκειται για τις ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι μάλλον οι συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να το διευκρινίσετε αυτό. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να το ελέγξω το συγκεκριμένο σημείο, Πρόεδρε. Αλλά νομίζω πως η συζήτηση που έγινε εδώ έδειξε πως υπάρχει μια μεγάλη γκάμα απόψεων, η οποία επιχείται και στις τροπολογίες που κατέθηκαν. Και ναι, Κριστίδη, έχει δίκιο σε αυτό που είπε ότι δηλαδή ενδεχομένω θα είναι δύσκολο να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τι διάφορε απόψει, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση και να φτάσουμε σε κοινέ προτάσει, οι οποίε θα συγκεντρώσουν δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη των ε, πολιτικών ομάδων ε, στην ε, Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα, Πρόεδρε, θα το ελέγξω και θα επανέλθω. Ευχαριστούμε τους πάντες, λέω ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τους Γερμανείς. Αύριο στις 9 το πρωί θα συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Πέρα στις συνεδρίες.